Ευχαριστώ συνάδελφοι που ήρθατε στην ώρα σας. Ξεκινάμε νωρίτερα όπως σας είπαμε. Σιγά σιγά μπορεί να αρχίσουμε να ξεκινάμε και στην ώρα μας. Χαίρομαι ιδιαίτερος και είναι ιδιαίτερη τιμή που μπορώ να καλωσορίσω τους τέσσερις εκλεκτούς και έγκριτους πανελίστες μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η στρατιωτικοποίηση του εύξηνου πόντου. Και βεβαίως ξεκινούμε ε, υπό την αιγίδα των σωμάτων της, ε, και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγγνώμη, και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο κύριος Στανισλάβ Τσεκουέρου. ο οποίος είναι fellow professor στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. ISS και θα μας κάνει μια παρουσίαση για αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε επίσης ε, εκπρόσωπο της Αμερικανικής Ναυτικής Δύναμης Επίσης έχουμε μαζί μας και τον κύριο Πατούκου Αντιπρόεδρο του Ατλαντικού Συμβουλίου της Γεωργίας και επίσης εκπρόσωπος του McCain Institute, πολύ γνωστό Ινστιτούτο. Και τέλος, αλλά οπωσδήποτε όχι ελάσσονος σημασίας, ο κύριος Ριβανμπάρη, ο Κώστα, ερευνητής, research Fellow ενός εξαιρετικά γνωστού πολωνικού πανεπιστημίου, του καλύτερου από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και ε, ασχολείται ε, με θέματα διεθνούς έρευνας για το πανεπιστήμιο που μόλις ανέφερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Το θέμα της ασφάλειας ε, στην λεκάνη του ευξήνου Πόντου είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας και μεταξύ των θεμάτων που εξακολουθούν να είναι μείζωνο σημασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε πέρσι και την ε, εξαιρετική έκθεση του Ιωάννου Μιρσέα Πάσκου για το θέμα αυτό Παρακαλώ πολύ να λείψουν τα πηγαδάκια και να μιλάτε χαμηλόφωνα γιατί μας ενοχλείτε, παρατηρεί η Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν την έκθεση Πάσκου ε, η οποία ανέλαβε ιδιαίτερη σημασία και διάσταση μετά από την παράνομη εισβολή και εξίσου παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ρωσία. Το θέμα αυτό λοιπόν παραμένει υψηλής προτεραιότητας. Η Μαύρη Θάλασσα και η γενικότερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι από τις πιο ευαίσθητες περιοχές ε, που μας ε, αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχουμε προβλέψει σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες συζήτησης. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, πανελίστες να πάρουν το λόγο ε, ε, με μία πρώτη εισήγηση 15 λεπτή και μετά να έχουμε ερωτήσεις και ένα δεύτερο γύρο μετά από σας, δηλαδή να εμπλακούν και τα μέλη στη συζήτηση έτσι ώστε να γίνει πιο επικοδομητική και πιο εμπλουτιστική. Βεβαίως, Δεν θα σας πάρουμε το κεφάλι αν μιλήσετε λίγο παραπάνω από τα 15 λεπτά, αλλά παρακαλώ να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Στανισλάβ Σεκέρο θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου έχετε απευθύνει. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον ε, τέτοιου ε, έγκριτου κοινού για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Παρακολουθώ καθημερινά την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και βεβαίως προκύπτει από αυτή την παρακολούθηση ότι η Ρωσία είναι ο κύριος παίχτης στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω να αποκαλύψω διάφορες φάσεις της ρωσικής στρατιωτικοποίησης στην περιοχή. Θα σας παρουσιάσω επίσης τις απειλές οι οποίες προκύπτουν από την ρωσική παρουσία στην περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για, άλλους, ε, ε, για άλλες περιφέρειες και περιοχές του κόσμου <clears throat> και ενδεχομένως στο τελευταίο τμήμα της παρέμβασής μου θα ασχοληθώ με κάποιες λύσεις τις οποίες ε, θα μπορούσα να δώσω ως ενδεχόμενα, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπισης της απειλής αυτής. Όταν μιλάμε για στατικοποίηση, συνήθως αναφερόμαστε σε κλασικούς όρους ανάπτυξης ε, ε, στρατιωτικών βάσεων, στρατιωτικές ασκήσεις κλπ. Ισχύει αυτό και τα είδαμε αυτά να συμβαίνουν τα τελευταία πέντε χρόνια στη λεκάνη του Ευξήνου Πόντου, αλλά δεν σταματάει εκεί η ιστορία. Η στρατιωτικοποίηση από την πλευρά της Ρωσίας είναι πολύ, μια διαδικασία πολύ πιο περίπλοκη ε, και ξεκινάει η περιπλοκότητα από το γεγονός ότι ε, η στρατιωτικοποίηση έχει πολλές διαστάσεις και πολλούς στόχους. Μπορώ να πω ότι η ρωσική στρατιοποίηση έχει πολλούς στόχους. Εννοώ ότι καλύπτει εγχώριους στόχους, αλλά και στόχους που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Η στρατιωτικοποίηση λοιπόν σχηματοποιείται ε, μέσα από στρατιωτικοποίηση του πολιτικού λόγου, ε, της πατριωτικής εκπαίδευσης στην Ρωσία, ε, των κοινωνικών συμβάσεων ακόμα και στατικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Εάν δείτε τώρα την εγχώρια πλευρά, τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται, η στατικοποίηση βεβαίως ε, μέσω του πολιτικού λόγου ε, έτσι ώστε να αφαιρέσει την δυνατότητα αφηγήματος από την αντιπολίτευση ε, με την έννοια που ε, ε, οι άνθρωποι οι οποίοι εντός της Ρωσίας θεωρούν ότι δεν είναι σωστοί, αντιτίθενται στην προσάρτηση της Κρυμαίας, θεωρούνται ανοιχτά ε, ως πολέμη της ε, χώρας ε, και επομένως θεωρείται ότι παίρνουν θέση σε αυτήν την υποτιθέμενη διαμάχη και χρησιμοποιείται επίσης για να αυξήσει την λαοφιλία και την δημοφιλία της κυβέρνησης η οποία αναφέρεται βεβαίως πάντα σε στρατιωτικές επιτυχίες. Ταυτόχρονα η στρατιωτικοποίηση κρίση έχει αντίκτυπο στις κοινωνικές ε, ε, συμβάσεις. Πριν η κυβέρνηση ε, ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να εγγυηθεί ας πούμε την ευμάρεια των ανθρώπων αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν λόγω της στρατιωτικοποίησης. Ο κόσμος απατηλά ε, τρέφεται ε, ή του παρουσιάζονται ε, νίκες οι οποίες παρουσιάζονται από τους πολιτικούς. Επίσης έχουμε την στερεωτική εθνικιστική εκπαίδευση με διτή μορφή ή πολυσχηδή μορφή Έχουμε τους νέους που ενθαρρύνονται όλο και περισσότερο να αγοράζουν συγκεκριμένα t-shirt ε, ή ε, διάφορα ε, προϊόντα μαζικής κατανάλωσης που έχουν πάνω στρατιωτικά σλόγγαν ή τέλος πάντων εικόνες με τα όπλα τα οποία παράγει η Ρωσία ή ακόμα υπάρχουν και κάποια προγράμματα πατριωτικής εκπαίδευσης που ήταν και παλιότερα παράδοση στην Ρωσία. Ε, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ακόμα και στρατιωτικούς οι οποίοι πηγαίνουν στα σχολεία ε, για να εκπαιδεύσουν ε, τα παιδιά. Ένα άλλο στοιχείο ή μια άλλη πτυχή της στρατιωτικοποίησης είναι μια περαιτέρω πτυχή στρατιωτικοποίησης, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτήν ενδεχομένως αργότερα. Έχει την οικονομική διάσταση της στρατιωτικοποίησης. Η στρατιωτικοποίηση επίσης έχει και μια εξαιρετική, συγγνώμη, εξωτερική διάσταση επίσης, καθότι υποστηρίζει την ε, Ρωσία στα πλαίσια μιας ισχυρής εξωτερικής ε, πολιτικής, ε, διότι εξυπηρετεί το στόχο της εξωτερικής πολιτικής όχι δια της πυθούς ή της έλξης, αλλά δια της αποτροπής διότι η Ρωσία παραδοσιακά θέλει να ονομάζεται ισχυρή δύναμη hard power. Ε, τέτοιου είδους εξωτερική πολιτική σημαίνει ότι το κατόφλι χρήσης ε, ε, ισχύ ισχύως έναν των γειτόνων έχει κατεβεί πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, η στερεωτικοποίηση οδηγεί σε αποσταθεροποίηση των ισορροπιών στην λεκάνη του ευξήνου πόντου. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια συστημική προσπάθεια αλλαγής της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή αυτή. Ε, η στρατιωτικοποίηση της ε, ε, εξωτερικής πολιτικής και η χρήση στρατιωτικών εκφάνσεων στην εξωτερική πολιτική οδηγεί την Ρωσία στο να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική ε, εξουσία ή ισχύ που έχει έτσι ώστε να ασκήσει βέτο σε κάποιες αποφάσεις που αφορούν την περιοχή. Αυτό βεβαίως μπορεί να αποσταθεροποιήσει, να αποσταθεροποιήσει ακόμα και να δυναμητήσει την ε, ε, γενική ισορροπία των γειτονικών χωρών και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να έχει σταθερούς ε, όμορους ε, ε, γείτονες. Η στρατιωτικοποίηση επίσης προωθεί την σοβιετική δύναμη προς τον Νότο. Είπα προηγουμένως ότι η στετικοποίηση είναι πολυσχηδής αλλά και πολλαπλών διαστάσεων. Εννοώ ότι αναλύοντας το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να μιλάμε μονάχα και να αναφερόμαστε στα καθαρά στρατιωτικά στοιχεία. Γιατί η Ρωσία έχει ε, κάνει την επιλογή πολυφασματικού πολέμου. Σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ε, και μη συμβατικά και λιγότερο ορατά εργαλεία για να επιτύχει τους στόχους της. Δεν μπορώ να μπω σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες ε, ε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, γνωρίζουν πολύ καλύτερα το θέμα και μπορούν να αναφερθούν σε αυτό. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέποντας την στρατιωτικοποίηση της λεκάνης του Ευξήνου Πόντου πέρα από την στρατιωτικοποίηση των νέων δογμάτων θα πρέπει να δούμε πώ. Ε, αυτό ε, μπορεί, αυτή η στρατικοποίηση μπορεί να συνδυαστεί ε, και με το κυβερνοέγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ξεκινήσω από τα πιο προφανή. Η στρατιωτικοποίηση σκοτώνει ανθρώπους. Έχουμε πάνω από 10.000 ε, ε, Ουκρανούς που έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της ε, εισβολής και της επίθεσης της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Επίσης, η στρατικοποίηση δημιουργεί πρόβλημα ε, στις αεροπορικές ε, ε, μεταφορές και καμιά φορά σκοτώνει και ανθρώπους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην υπορωσικό έλεγχο περιφέρεια της Ντομπάσα είχαμε την κατάρριψη του επιβατηγού αεροπλάνου. επίσης, ε, γνωρίζουμε ότι ε, χρησιμοποιείται ε, η παρέμβαση της Κρυμαίας έτσι ώστε να δημιουργήσει, να εντείνει ακόμα περισσότερο και την κρίση στην Συρία. Δημιουργεί αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, απειλούνται όχι μόνο άμεσα ε, χώρες όπως η Ρουμανία ας πούμε, ε, αλλά ε, υπάρχουν και απειλές για άλλες πιο μακρινές περιοχές μέσω των βαλιστικών πυράβλων Εβραίους Βελληνικούς. Η πατριωτική εκπαίδευση εντός της Ρωσίας, κατά την άποψή μου όμως, είναι αυτή η οποία ε, θα ε, δώσει ένα αποτέλεσμα, θα δώσει ως αποτέλεσμα μία ε, στην καλύτερη περίπτωση πιο αδιάφορη, στην χειρότερη περίπτωση πολύ πιο επιθετική γενιά Ρώσων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μυριάδα προβλημάτων που προκύπτουν από την ρωσική στρατιωτικοποίηση. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ε, θα αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα σταθή πολιτική ελίτ στην ε, Ρωσία. Δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Τη μία μέρα θα βλέπεις έναν άνθρωπο, την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει πια. Ε, ε θα αντιμετωπιστεί επίσης ενδεχομένως το φαινόμενο μιας ε, στασιμότητας ε, στην ρωσική οικονομία, ταυτόχρονα με γυράσκοντα πληθυσμό και, όπως έλεγα και προηγουμένως, μια ιδιαίτερα διάφορη ή ακόμα και επιθετική νέα γενιά για το μέλλον και δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα, δεν θα, δεν θα έχετε στο Κρεμλίνο ε, έναν εταίρο που θα, είναι, που θα δίνει τη δυνατότητα για στενή, ε, αξιόπιστη, καλή οικοδομητική συνεργασία. Θα πρέπει επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτή τη ρωσική πρόκληση και δυστυχώς δεν υπάρχουν ε, θαυματουργές Πολλά στοιχεία είναι σημαντικά για την επιτυχία της ρωσικής, διορθώνω, της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με τη Ρωσία. Πρώτον, η ενότης. Έστω και αν αυτό είναι απολύτως ε, αυτονόητο, πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Ενότηση απέναντι στη Ρωσία. Ε, έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και είναι σημαντική. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι διαιρεμένη, τότε ε, η Ρωσία θα έχει, το Κρεμλίνο θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να επιτύχει τους στόχους του. Ε, δεν μπορούν να αρθούν και δεν πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις εάν η Ρωσία δεν αποδεχτεί όλους τους όρους που είχατε εκ των προτέρων θέσει. και ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μακροχρόνια επένδυση για τους ε, ανατολικούς ε, γείτονες. Είπαμε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας είναι πολυφασματικός. Αυτό το ευρύ φάσμα λοιπόν ε, ε, πολεμικής ε, δύναμης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από, ένα ευραίος, από μια ευραίος φάσματος ανταπόκριση και θα πρέπει λοιπόν με αυτό τον τρόπο να απαντήσετε στην ρωσική απειλή αν θέλετε να είστε αποτελεσματικοί. Η Ρωσία προκαλεί πρόβλημα διαταράσει τις εμπορικές ισορροπίες ισορροπίες και συμφωνίες στην περιφέρεια του, του, του Ευξήνου Πόντου. Επομένως, ε, θα πρέπει να βοηθηθούν οι εταίροι της ανατολικής εταιρικής ε, ε, σχέσης. Ε, είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία που έχετε να ξανασκεφτείτε και κάποια εργαλεία τα οποία καλύτερα θα βοηθήσουν τους γείτονες και θα δώσουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε, πολλαπλούς, σε πολλαπλές απειλές. Εσείς επίσης θα πρέπει να προσπαθήσετε να δείξετε ε, ε, ε, γέφυρες στην, προς την κοινωνία της Ρωσίας. Θα υπάρξουν δυσκολίες οπωσδήποτε, θα υπάρξουν αποτυχίες γιατί δεν θέλει τέτοιες εμπλοκές η Ρωσία. Ωστόσο, ενδεχομένως θα βελτιωθούν μελλοντικά οι σχέσεις με τη Ρωσία σε αντιπαράθεση με αυτήν την γενιά αδιάφορων και εχθρικών ατόμων που προσπαθεί να οικοδομήσει η Ρωσία. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στίβεν Χόρο, πλωτάρχης, ο οποίος ε, συμμετέχει σε εργασίες του Ατλαντικού Συμβουλίου, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ στρατηγική, λέει ο πλήρχος. Ε, παλιά ήταν συγκεκριμένα που συζητούσαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε τη συμμαχία αυτή για να αναπτύσσουμε ε, συζητήσεις για τα θέματα για να συνεχίσουμε δεν συμμετέχω πλέον στο Ατλαντικό Συμβούλιο είμαι εδώ ε, ως ιδιώτης και εκφράζω τις δικές μου απόψεις καμία επίσημη άποψη του Υπουργείου Αμήνης στον ΗΠΑ Έχοντας δηλώσει αυτό, ας ασχοληθώ με το θέμα της στατικοποίησης στον εύξηνο πόντο. στο έγγραφό μου αναφέρομαι στο τοικικό περιβάλλον και τη στατικοποίηση, αλλά πιο σημαντικά στην αύξηση της αντιπαράθεσης με την Ρωσία και να αναφερθώ σε κάποιες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια θα ήθελα, από όταν συνεγράφει το έγγραφό μου και ποια θα στρατηγική και η πολιτική βάσει των συστάσεών μας για το ΝΑΤΟ, για τη Δύση, τεχνικές πτυχές. Κάποιες εντάσσονται στη στατικοποίηση από τις συστάσεις. Θέλουμε αυξημένη παρουσία και αύξηση των ασκήσεων. Αυτές τις συστάσεις θα ήθελα να τις εξετάσουμε μαζί με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο. Βεβαίως δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες στις απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις. Θα αναφέρω διπλωματικές ε, πτυχές, οικονομικές πτυχές, ενεργειακές πτυχές. από τον Οκτώβριο του 2016 στο συζητήσαμε στο Τελικό Συμβούλιο το στατικό περιβάλλον τευξίνου πόντου. Εξετάσαμε το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, την αύξηση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσεως. Τώρα, αν η Δύση θεωρείται από τη Ρωσία ότι είναι η ΕΠΑ, ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ΝΑΤΟ, ή γενικότερα η Δύση, πάντως υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Το σημείο καμπής στην αύξηση της διαφοράς ε, είχε σαν επίκεντρο τον εύξηνο πόντο, οι αλλαγές στην Ουκρανία, η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, αυτή καθε αυτή σαν πράξη και ακόλουθες δράσεις αύξησαν τη στατικοποίηση. Και αυτή η ταχεία κλιμάκωση συνέβη σε μια περιοχή όπου υπήρχαν διάφορα σημεία προστριβής με παρατεταμένες συγκρούσεις στον Εύξηνο Πόντο και στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Ευξηνού Πόντου. Η προσάρτηση της Κρυμαίας ακολουθήθηκε από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας υπό την, ε, την ηγεσία της Ρωσίας. Στην Κρυμαία η προσάρτηση έγινε σχετικά γρήγορα και σχετικά ανέμακτα και καλύφθη μετά με πολιτική κάλυψη δημοψηφίσματος το γεγονός. Αμέσως μετά, σχεδόν, η Ρωσία μετακίνησε στρατιωτικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στην κατεχόμενη αυτή Χερσόνησο και ο στόλος ήταν σεβαστού πολύ ε, της Μαύρης Θάλασσας αλλά μετά την προσάρτηση έφερε ε, πυράβλους εδάφους αέρα και ε, πυράβλους κρούς έτσι αυξήθηκε η δυνατότητα της Ρωσίας να περιορίζει χώρους, να ελέγχει χώρους, εναέριους, χερσαίους, να καλύπτει τον μισό εύξηνο πόντο. Επίσης, συνέχισε τον εξυγχρονισμό του στόλου του ευξήνου πόντου, βελτίωσε την κατηγορία των υποβρυχίων με κινητές δίζελ, ε, που είναι εξοπλισμένα πυραυλικά συστήματα. Επίσης νέα συστήματα φρεγατών με προωθημένα συστήματα πυραυλικά. Δεν είναι μόνο πύραυλοι ε, θάλασσας-θάλασσας αντί ε, κατά των σκαφών, αλλά είναι πύραυλοι κρούζ οι οποίοι μπορούν να επιτεθούν καθιοδήποτε, οδήποτε στόχους σε μια περιφέρεια, σε μια εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το βεληνικές τους από το 2010 είχαν προγραμματίσει τις κινήσεις τους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προωθεί την τεχνολογία εχμής τη στρατιωτική στην περιοχή και συγχρόνω παίρνει θέση αντιπαράθεση με τη Δύση. Υπήρχαν προκαθορισμένα σχέδια για την αύξηση του στόλου και τον συγχρονισμό αυτού τον εύξηνο πόντο. Άρα είχε σκοπό να στατικοποιήσει τον εύξηνο πόντο η Ρωσία από παλιά. Πρέπει να τονίσουμε τι έγινε στον ένα χρόνο από όταν δημοσιεύθηκε το έγγραφό μου. Στο έγγραφό μου ανέφερα τι πρώτε παραδόσει των υποβρυχίων και των φρεγατών. Και τώρα τα υποβρύχια του εύξηνου πόντου τελευταία εβδομάδα απέπλευσαν από τον εύξηνο πόντο και πήγαν στην Ανατολική Μεσόγειο και ε, έστειλαν πυράβλους ε, θαλάσσις εδάφους ε, στη Συρία. Αυτή η στατικοποίηση του ευξήνου πόντου έχει συνέπειες. Αυτές που ανέφερα που ξεπερνούν τα στενά όρια της περιοχής και πέρα από τις χώρες που είναι γύρω από τον πόντο. Στο έγγραφο ήθελα να τονίσω σημεία για τις στρατηγικές απαντήσεις θα βρει το ΝΑΤΟ, που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής. Στο επίκεντρο ήταν το ΝΑΤΟ του εγγράφου και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν και ο στόχο των συστάσεων. Αν το πρόβλημα είναι η στατικοποίηση του ευξήνου πόντου, θεωρώ ότι η λύση πρέπει να επικεντρωθεί επί της πλέον επιτυχού στρατιωτική συμμαχία που υπήρξε ποτέ. Το ΝΑΤΟ έχει τη στρατιωτική δομή την κατάλληλη, ούτω ώστε να είναι το κομβικό σημείο δυτικοευρωπαϊκή απάντηση στην επιθετικότητα και στατικοποίηση τη Ρωσία στην περιοχή. Τι έκανα λοιπόν, συνέστησα αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και ασκήσεις. Θαλάσσια παρουσία κατά περιόδους, τα δυτικά κράτη που δεν έχουν ακτές στον εύξηνο πόντο είναι περιορισμένα στον αριθμό, ε, σε χωρητικότητα πλοίων και το χρόνο που μπορούν να βρίσκονται στον εύξηνο πόντο, αλλά με κυκλική αναλλαγή μπορούν να παρίστανται. Και κυκλική ενέργεια παρουσία με κυκλική αναλλαγή που εκεί δεν έχουμε τόσους περιορισμούς. Επίσης παρουσία επί εδάφους με χερσαίες ασκήσεις, βελτίωση των τοπικών δομών για τις στατιωτικές δυνάμεις της χερσαίας στην περιοχή ε, του Ευξήνου Πόντου. Όπως προανέφερα, τα είδα όλα αυτά από τη σκοπιά του ΝΑΤΟ. Όμως μπορούσαν να συμμετέχουν και περιφερειακοί εταίροι που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Θα ήταν σημαντική για την προσπάθεια. Έκτοτε είχαμε και άλλες εξελίξεις και στη Δύση. Αυτή την εβδομάδα η πολυεθνής μονάδα η Νοτιοανατολικής Ευρώπης εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία. Είναι ε, αμυντικό σύστημα που εγκαταστήσαμε κατά των βαλιστικών πυράβλων και είχαμε την, άμυνα, την άσκηση Falcon 2017 με F-16 πορτογαλικά που απογειωθήκαν από τη Ρουμανία και είχαμε και χερσές ασκήσεις Ατλαντική αποφασιστικότητα, τον τίτλο Atlantic Determination στην Βουλγαρία, 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια, 40.000 στρατιώτες από 22 χώρες συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση. Κατά την άποψή μου όλα αυτά είναι καλά και άγια. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ε, δημιουργείται συλλογική άμυνα, τι το και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Επισημαίνω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που είναι άκρο αξιόπιστα υπό την ηγεσία των μελών εκείνων του, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ που έχουν ακτές στην, στον αλλά και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ ε, μεγιστοποιούν τις προσπάθειες και συμμετέχουν με κυκλική αναλλαγή στην παρουσία ε, στον Εύξηνο Πόντο. Ακόμα και αν δεν είναι υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, ακόμα και με εθνική σημαία μπορεί να γίνει συντονισμός ε, στο κέντρο επιχειρήσεων και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι στη Δύση. Μετά η αποστολή δημιουργίας αμυντικής δυνατότητας και για τις χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αυτοί μπορεί να συμμετέχουν διμερό, πολυμερό, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων. Μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτοί οι εταίροι δεν οίκουν στο ΝΑΤΟ, σε εκδηλώσεις του ΝΑΤΟ και σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Αν γίνει σωστά, δημιουργείται δυναμικότητα, αυξάνονται δυνατότητες και ενισχύονται οι διασυνδέσεις, έχουμε περιβάλλον ασφαλείας και αν κινηθούμε σωστά μπορούμε να αποφύγουμε τις προκλήσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, την πρόκληση, είναι σημαντικό να αφήνουμε και την πόρτα ανοιχτή για τη Ρωσία, να επιτρέψουμε στη Ρωσία να δείξει ότι είναι υπεύθυνο εταίρος στο διεθνές προσκήνιο. Η το ΝΑΦΟΡ του Ευξήνου Πόντου παλιά συμπεριλάμβανε τη Ρωσία και άλλες περιφερειακές χώρες. Αυτό ανεστάλλει με τέτοια παρόμοια δυνατότητα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για τη συμμετοχή της Ρωσίας εκ νέου, να μπορεί να είναι ξανά εταίρος σε κάποιες διεθνείς προσπάθειες για την ασφάλεια παρά να είναι σε θέση αντιπαράθεσης συνεχώς. Κλείνοντας, να πω ότι είπε ο Γενικό Γραμματέα, ο κ. Στότελμπεργκ, στην Κραϊόβα, στην, στην στη Ρουμα... μάλλον στην Κραϊόβα, στη Ρουμανία, είπε την περασμένη εβδομάδα, δεν είμαστε απειλή για τη Ρωσία, χρειαζόμαστε διάλογο όμω από ισχυρή θέση Άμυνα και αποθάρρυνση τέλο παράθεση. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω. Προσβλέπω στη συνέχεια των συζητήσεων. Θέλω να ακούσω σχόλια, ερωτήσεις και τη συνέχεια της συζητήσεως. Ευχαριστώ. Ήταν η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως και μπορέσαμε να τα ακούσουμε αυτά που αναφέρατε. Ε, όλη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του κ. Στότερμπεργκ, πολύ ισχυρά τα λόγια του. Ε, ο κ. Μπάτο Κουτέλια μπορεί να λάβει το λόγο τώρα. Αντιπρόεδρος του Τατατικού Συμβουλίου της, ε, και είναι και μέλος του Ινστιτούτου Μακέινς. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για αυτό το στρατηγικά δύσκολο θέμα ε, το οποίο έχει ε, σημαντική επιρροή στην ασφάλεια της ασφάλειας στην ευρωατλαντική περιοχή. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω κάποια από τα σημαντικά πράγματα τα οποία είπαν οι προηγούμενοι μελητές και με τους οποίους συμφωνώ απόλυτα. Βλέποντας όμως τη γενικότερη εικόνα θα πρέπει να θυμόμαστε το γενικότερο ε, πλαίσιο της ευρωτατικής ε, ασφάλειας ε, και τις εξελίξεις που παρατηρούνται στον έξινο πόντο. Όσον αφορά λοιπόν την ε, συγκεκριμένη ε, περιοχή, έχουμε ε, το πλαίσιο ειρήνης και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει μονάχα βασικά στοιχεία της διαμάχης με τη Ρωσία ε, έχουμε ε, την Ρωσία που προσπαθεί να αλλάξει την, ε, το status quo μετά τον ψυχρό πόλεμο. Έχουμε την, τη Μαύρη Θάλασσα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης. Για να βρεθεί λοιπόν μια νέα ισορροπία στην Μαύρη Θάλασσα θα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να θυμόμαστε το μη αναστρέψιμο της όλης διαδικασίας, ε, το οποίο ε, μπορεί να συμβεί μονάχα με μια στρατηγική δυτική προσέγγιση. Όπως γνωρίζουμε, ε, λοιπόν, η Ρωσία ε, ισχυρίζεται ότι η βασική αντίπαλη είναι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα πρέπει να θυμούμαστε ότι για αυτούς τους σκοπούς λοιπόν η Μαύρη Θάλασσα έχει, πάρα πολύ έχει μεγάλη σημασία για τη Ρωσία για να δείξει τη δύναμή της προς Ανατολάς αλλά και προς τις νότιες περιοχές της Ευρώπης. Αυτή ε, τη στιγμή η ανάπτυξη στην περιοχή είναι ε, σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση, ε, το οποίο είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό με βάση τις μεθόδους αλλά και τις συνέπειες. Μιλώντας ε, λοιπόν για τη στρατηγική προσέγγιση την οποία προσπαθεί να ακολουθήσει η Ρωσία, η βασική στόχη είναι να σταματήσει ε, την ε, δυτική δημοκρατική εξέλιξη διότι αυτήν τη θεωρεί ως απειλή. Θέλει να κρατήσει λοιπόν την κατάσταση του ψυχρού πολέμου και θέλει να δημιουργήσει βέβαια και ζώνες επιρροής επίσης ε, θέλει να ε, πνίξει τους, ε, τους ενεργειακούς, τις ενεργειακές οδούς προς προορισμούς που δεν συμφέρουν την Ρωσία. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ενεργειακές κρίσεις και παράλληλα βασικό στοιχείο είναι να δείξει ε, ότι ε, οι δημοκρατικές αξίες δεν συμφέρουν τους γειτονές της ε, και επίσης θέλει να υποστηρίξει ακροαριστερές ή ακροδεξιές παρατάξεις και κινήματα. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι θέλει να προκαλέσει την δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προπογάνδας σε διάφορους τομείς η στρατηγική αυτή είναι υβριδική και και γίνεται με έναν τρόπο προκαλώντας τις κόκκινες γραμμές. Ε, προσπαθεί δηλαδή ε, να ε, τις σμπρώξει και να δημιουργήσει νέες πραγματικότητες. Μετά την την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας ε, η Ρισαία προκάλεσε ε, τους διεθνείς θεσμούς όπως είναι για παράδειγμα ο ΙΕ και ο ΑΣΑ και με αυτόν τον τρόπο ο επόμενος στόχος που θα προκαλέσει η Ρωσία θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και ε, μέσα, μέσω αυτής της μεθόδους πολλοποίησης και κατάκτησης ε, και παραλύοντας την πολιτική ε, διαδικασία βλέπουμε ότι είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική. Έχουμε το πλοίο Μίστραλ, το οποίο ε, προσπάθησε να καταλάβει και ε, το οποίο ε, προκάλεσε αντιδράσεις από τον ΝΑΤΟ και τη δυτική κοινότητα, συνδυασμό στρατιωτικών ασκήσεων και στη συνέχεια η εισβολή σε ανεξάρτητες χώρες όπως έγινε στην Ουκρανία και στη Γεωργία όπως επίσης και ε, διαφορομαθήματα της Ρωσίας ότι αν δεν ελέγχει την ε, παροχή μέσω της ε, Μαύρης Θάλασσας τότε θα είναι αδύνατο να επιτύχει τους στόχους της πέραν του απλά να καταλάβει κάποιες περιοχές. Στη ε, γεωργία λοιπόν ε, πέρα από τις κατηλημένες ε, περιοχές. Το φαινόμενο αυτό καταλήφθηκε διότι οι ΙΠΑ χρησιμοποίησαν στρατιωτική διπλωματία και επίσης δεν μπόρεσαν να προωθήσουν τους στόχους τους. Ένα άλλο σημαντικό ε, στοιχείο αυτών των πολεμικών παιχνιδιών της ε, Ρωσίας είναι ένα πλαίσιο το οποίο αναφέρθηκε, το οποίο είναι η, πρόσβαση, η άρνηση πρόσβασης ε, ε, αυτό συνδυάζεται και από αερός αποκλεισμούς με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ε, περιοχές, ε, αποκλεισμένες περιοχές και άμα εξετάσουμε λοιπόν τα συστήματα της Ρωσίας, τα αεροπορικά συστήματα της Ρωσίας, δημιουργείται μια τέτοια ζώνη απαγόρευσης. Υπάρχουν μόνο δύο κενά σε αυτό το σημείο ε, από τη μία η Γεωργία που, όπου έχει καταλάβει ήδη την Απχαζία και έχει ε, πυραυλικά συστήματα άμυνας και ένα άλλο στοιχείο αφορά την Τουρκία νότια της ε, Μαύρης Θάλασσας. Εκεί βλέπουμε όμως την εξέλιξη όπου ε, η Ρωσία προσπαθεί να πουλήσει το σύστημα S400 το οποίο, ε, η αγορά του οποίου μπορεί να ακυρωθεί με βάση τις τελευταίες ειδήσει, όμως παρόλα αυτά η Ρωσία προσπαθεί να επιβάλλει αυτά, αυτές τις τακτικές κινήσεις αυτό έγινε ορατό μετά από το 2008 όταν προσπάθησε ε, να αντιδράσει ε, στην Δύση. και στη συνέχεια η Ουκρανία και η ε, Γεωργία έγιναν θύματα της ρωσικής επιθετικότητας. Όσον αφορά τον αφοπλισμό, εκεί δημιουργείται μια βεβαιότητα και δημιουργεί ε, συμμαχίες ε, με ε, αυταρχικά καθεστώτα, το οποίο είναι κομμάτι της ρωσικής τακτικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, δημιουργούνται αυτές οι ζώνες από στρατιωτική άποψης, όμως από πολιτικής άποψης ε, προσπαθεί να ουδετεροποιήσει χώρες ή να προωθήσει την ιδέα μιας γκρίζας ζώνης ε, μέσω μη κρατικών παραγόντων. Και εδώ λοιπόν χρησιμοποιεί του τους στρατιώτες, τα πράσινα ανθρωπάκια, για το σκοπό αυτό και επίσης ο Πούτιν είναι ένα ε, στάνταρ πακέτο για τους αυταρχικούς ηγέτες ε, προσφέροντά τους ε, συνεργασία ε, και με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία προσπαθεί να επιβάλλει την δύναμή της ε, στις περιοχές ε, που θεωρούνται ότι αποτελούν στρατιωτικό συμφέρον, στρατιωτικό συμφέρον για, τις, για τη Ρωσία. Επίσης, η Μαύρη Θάλασσα προσφέρει πρόσβαση στη Μεσόγειο και στην Κασπία. Εδώ το βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τη μία στην, ε, στα ανατολικά της Ευρώπης λοιπόν θεωρείται η Ρωσία απειλή ενώ ε, στα δυτικά απειλή θεωρείται η τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά η Ρωσία προσπαθεί να χειρογηγήσει τα συγκεκριμένα ε, θέματα για να μεγαλώσει το χάσμα προς αυτή την αντιμετώπιση που υπάρχει. ενώ παράλληλα ε, προσπαθεί να ενισχύσει τις διαμάχες ε, στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσει περισσότερους ε, πρόσφυγες που θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Η καλή είδηση όσον αυτό είναι ότι η σύνοδος της Βαρσοβίας ήταν, ένα, ήταν πολύ σημαντική όσον αφορά την αντίληψη μιας κοινή απειλής και ε, είδαμε ε, ότι έχουμε αυτές τις δύο απειλές, το Ισλαμικό κράτος ε, και τη Ρωσία που περιλήφθησαν στην ίδια παράγραφο της ανακοίνωσης και έχουμε λοιπόν την δήλωση περί και μη κρατικών απειλών. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Επίσης η Μαύρη Θάλασσα περιλήφθηκε σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρθηκε συνολικά 8 φορές σε διάφορα κεφάλαια όσον αφορά τις ε, ε, περιφερειακές προσεγγίσεις ε, για τα ζητήματα ασφάλειας σε ευρωατλαντικό περιεχόμενο. Ένα άλλο πλαίσιο για να κατανοήσουμε την προσέγγιση της Ρωσίας προς αυτή την ε, περιοχή είναι, ε, αφορούν το ζήτημα των χωρών ε, στα ανατολικά του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ρωσία. Πρόκειται για σημαντικές χώρες τέρους, Σουηδία, Φιλανδία έχουμε εκεί πέρα και το ίδιο συμβαίνει και στη Μαύρη Θάλασσα. Όμως η περιοχή αυτή είναι λιγότερο ευέλετη διότι έχουμε ε, ισχυροί, ε, ε, χώρες που είναι ισχυρές από άποψης στρατιωτική και οικονομικής άποψης, ενώ από την άλλη έχουμε την Ουκρανία που θεωρείται ότι είναι πιο ευάλωτη στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την αυτοάμυνα αυτών των χωρών και αυτό αφορά την τον εξοπλισμό της Ουκρανίας ε, με όπλα, το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό για να αλλάξει τους στρατιωτικούς υπολογισμούς της Ρωσίας. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις ε, στην ε, συνέλευση του ΝΑΤΟ. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της τον ΙΠΑ, ο οποίος απέστειλε ισχυρά μηνύματα. Είχαμε την ε, παρουσία του ΝΑΤΟ στην ε, περιοχή, στη Ρουμανία. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν θα ήταν η περαιτέρω εξέλιξη ε, της της εμπορικής οδού μεταξύ ε, Ανατολής και Δύσης, το οποίο επίσης έχει στρατηγική σημασία διότι θα ανοίγει πρόσβαση στην Κασπία ε, και, στις, ε, και στους ενεργειακούς πόρους. Ταυτόχρονα όμως θα έδειχνε ότι πρόκειται για μια περιοχή προς που ενδιαφέρει τον πολιτισμένο δημοκρατικό κόσμο. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι σημαντικά. Πρώτον η ε, Κρυμαία ε, η οποία έδωσε περαιτέρω όρεξη στην Ρωσία ε, να επεκταθεί με περισσότερο στρατιωτικοποίηση των κατηλημένων περιοχών. Ε, ένα άλλο στοιχείο αφορά την Γεωργία και σε αυτή την περίπτωση η Γεωργία δεν είναι απλά μία μικρή χώρα που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας επιτυγχάνοντας τον ε, στρατηγικό στόχο και αλλάζοντας την ε, πολιτική της ε, γεωργίας, η Ρωσία θα μπορέσει να αρνηθεί πρόσβαση στην Κασπία και στη συνέχεια στην Κεντρική Ασία για το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα μπορούσε να αποστείλει η Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο οι κατηλημένες ε, περιοχές ε, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την ε, πολιτική της Ρωσίας και ιδιαίτερος η στρατιωτικοποίηση της Απχαζίας στη Γεωργία όπου η Ρωσία ήδη έχει εξοπλίσει περαιτέρω την, διάφορες βάσεις που υπάρχουν εκεί μεταξύ άλλων έχει ε, στείλει 130.000 στρατιώτες ε, στις περιοχές, ε, στις περιοχές όπως επίσης και λοιπό στρατιωτικό εξοπλισμό με αυτήν τη στρατιωτική παρουσία και με την πίεση που ασκεί στην ε, γεωργιανή κυβέρνηση προσπαθεί να απομακρύνει τη Γεωργία από την ενσωμάτωσή της ε, στο ΝΑΤΟ και να αποτρέψει αυτή την ιδέα δυτικοποίησης ε, στοχοποιώντας μέσω προπαγάνδας τις δυτικές αξίες. Επίσης απαιτείται ε, όχι μονάχα αποτροπή μέσω της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ ε, στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχουν όμως ε, συζητήσεις σχετικά με το αν θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε την στρατιωτικοποίηση της Ρωσίας μέσω ενίσχυσης του ΝΑΤΟ ή αν θα επιλέξουμε μια ισορροπία. Η δεύτερη λοιπόν εναλλακτική θα ήταν λαθασμένη όσον αφορά τη στρατηγική στη Μαύρη Θάλασσα διότι ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, οπισθοχώρηση της Ρωσίας, ε, θα μπορούσε, ε, θα απαιτούσε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά και επίσης περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη. Εν συμπεράσματι λοιπόν, να πω μερικά πράγματα ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δημοκρατική Κοινότητα, το ΝΑΤΟ ε, ε, δεν θα πρέπει να ε, λένε ότι θα πρέπει απλώς να ε, κάνουν διαχείριση της κρίσης. Αυτό θα ήταν λάθος. Ε, δεν θα ήταν σωστό επίσης να δημιουργηθεί ένα κενό το οποίο οπωσδήποτε θα καλύψει η Ρωσία και η ρωσική προπαγάνδα και επίσης δεν θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες εμπορικές ας πούμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα status κβο γιατί η τέτοιου είδους σταθεροποίηση, η κατάθεση ε, θα ξυπνήσουν ψυχροπολεμικές ε, μνήμες. Αυτά και περιμένω ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο ε, Ρίτβαν Μπάρι Ουρκώστα να πάρει το λόγο. Uh, Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ο κύριος Κουτέλια έκανε είπε δύο για την Κρυμαία και κατά κάποιο τρόπο ε, μας έδωσε, έτσι έκανε μια εισαγωγή σε αυτά που θέλω να πω εγώ για την Κρυμαία, για τη θάλασσα του Αζόφ ε, και, και ε, για τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν γύρω στα μέσα ε, του καλοκαιριού από ναυάρχους Ρώσους ε, οι οποίοι κοινοποίησαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την κατάσταση και τις βλέψεις που έχουν ε, όσον αφορά την λεκάνη του Ευξήνου Πόντου αλλά και πιο πέρα. Και θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη ρωσική πολιτική σε σχέση με την Ρωσία. Έχουμε δύο δεσπόζουσες δυνάμεις ε, στην Μαύρη Θάλασσα, τη Ρωσία και την Τουρκία. Αλλά η θέση της Τουρκίας είναι μάλλον ασαφής ε, για την ώρα. Αυτές είναι οι εικόνες από την, Σεβαστο... από την Σεβαστούπολη, από την οποία προέρχομαι άλλωστε. Είμαι γηγενής. Ε, φωτογραφίες του 2014 λοιπόν και βλέπετε την ε, απέλπιδα κατάσταση το, και την πλήρη καταστροφή του παράκτιου συστήματος ε, άμυνας. Αυτό που έχουμε τώρα όμως Ζητούμε συγγνώμη, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα από τη μεριά του ομιλητή. Yeah. Can you go back? Yes. Click, please. Yes, I would like to show what kind of situation right now. Yeah. With this. So it's like a, the more the main picture η κύρια εικόνα στρατικοποίησης ε, της ε, Κρυμαίας από την ε, Ρωσία, μάλλον οι εικόνες που σας δείχνω, ακριβώς αποδεικνύουν πόσο, πόσο λειτουργεί το σύστημα. Όμως τώρα όλα έχουν εξυγχρονιστεί, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γραμμή άμυνας της Κρυμαίας. Ναι, ήθελα να σας δείξω σε αντιπαράθεση τις εικόνες του πριν,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 Ε, θα πω δύο λόγια για να δείξω γιατί η Κρυμαία είναι σημαντική για την ε, ε, Ρωσία. Για λόγους ιστορικούς πρώτα απ' όλα. Η Ρωσία χρησιμοποίησε την Κρυμαία έτσι ώστε να κάνει επίδειξη δύναμης Στην πρώτη προσάρτηση 200 χρόνια πριν ε, χρησιμοποιήθηκε η Κρυμαία έτσι ώστε ε, να δείξει η Ρωσία ότι έχει μεγάλη ε, δύναμη προς όλες τις κατευθύνσεις όπως είχε κάνει παλιότερα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κρυμαία άλλωστε είναι το μόνο σημείο στην, στον εύξηνο πόνο που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο όλης της λεκάνης του Ευξήνου Πόντου. Όσον αφορά την Ουκρανία, επίσης είναι πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Οι νότιες ε, περιφέρειες, ε, στον ε, οι ρωσόφωνες περιοχές, τις οποίες γνωρίζουμε, και επομένως ε, η ε, στρατικοποίηση της ε, Κρυμαίας ήταν πολύ σημαντική και για τους Ουκρανούς και αυτό το κατάλαβαν οι Ρώσοι. Και γι' αυτό ακριβώς έβαλαν στόχο την Κρυμαία. Από την προσάρτηση και μετά Α το πούμε πολύ απλά μάλλον από παλιότερο να ξεκινήσουμε, Στον, ε, στην περίοδο του ε, ψυχρού πολέμου τα πράγματα ήταν ε, διαφορετικά, ήταν μια ενιαία περιφέρεια. Τώρα όμως η Ρωσία την διαμέλισε γιατί ακριβώς είχε πρόβλημα με τους τάταρους της Κρυμαίας. Υπήρχαν και διάφοροι στρατιωτικοί σχηματισμοί στην ε, περιοχή αυτή και αυτό αποτέλεσε ένα σημείο σύγκρουσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση με την προσάρτηση είναι ότι στην ουσία η Ρωσία πλέον κατέχει ε, πλήρως την ακτογραμμή ε, της ε, Μαύρης Θάλασσας. Πράγμα πολύ σημαντικό από στρατηγική άποψη. Και ένα άλλο στοιχείο αφορά την Αζωφική θάλασσα, τη θάλασσα του Αζόφ. Για, διότι η Ουκρανία δεν έχει πλέον καμία στρατιωτική δυνατότητα για τη θάλασσα αυτή. Γιατί αν θέλει κανείς να ενισχύσει στρατιωτικά ε, τον ε, Ουκρανικό στόλο στη θάλασσα, αυτή ε, θα πρέπει να περάσει από τα στενά του Κέλτα. Αλλά τώρα πια η Ρωσία, όταν θα έχει ολοκληρωθεί μάλλον η σταθερή σύζευξη από την πλευρά της Ρωσίας, τότε και αυτό θα είναι δύσκολο. Ποιες είναι οι δυνατότητες κανάλι ε, από την Βόρεια Κρυμαία μέχρι τη θάλασσα του Αζόφ. Ε, δεύτερη δυνατότητα ε, είναι η χρήση μικρών σκαφών, λεγόμενος μοσκίτοφλι. Μικρά ευέλικτα σκάφη, τα οποία να μπορούν να κινούνται στην ακτογραμμή ένα είδος ε, ε, άμυνας της ακτογραμμής ας πούμε. Ωστόσο αυτό είναι δύσκολα επιτεύξιμο διότι έστω και αν ε, τα ονομάζουμε σκάφη κουνούπια, πολύ μικρά σκάφια, παρόλα αυτά είναι σκάφη τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παραδοθούν. Και αυτό δεν είναι προφανές στην Ουκρανία και πώς θα φτάσουν ε, ε, δυνάμεις ενίσχυσης, στρατιωτικής ενίσχυσης ε, της θάλασσας του Αζόφ. Yeah, yeah, it's better. Κατά τη διάρκεια της ε, ύπαρξης Σοβιετικής Ένωσης ε, η στρατιωτική ε, παρουσία ήταν στην Κρυμαία 70.000. Τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη παρουσίαση. Δεν, μάλλον δεν έχουμε συγκρίσιμη παρουσίαση, αλλά πάντως, παρουσία, αλλά πάντως έχουμε αυξημένη ε, στρατιωτική παρουσία που προσεγγίζει την παρουσία ε, της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης. Το βέβαιο είναι ότι η Ρωσία θέλει να επικεντρωθεί σε ε, υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. High-tech technology. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ να δούμε, ας πούμε, ότι η Ρωσία, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, έχει δημιουργήσει νέο ε, σύστημα ε, ελέγχου του συνόλου του ευξήνου πόντου, έτσι ώστε ο ευξήνος πόντος να μην χρησιμοποιηθεί μονάχα σαν προμαχώνας, αλλά και σαν ε, προωθημένη θέση. Αυτή η κατάσταση εδώ που βλέπετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρουμε το θέμα της γέφυρας του Κέλους, αλλά κανείς δεν λέει τι γίνεται με ένα άλλο σημείο. Έχουμε ε, τον θερμοπαραγωγικό σταθμό της ε, ε, Σεβαστοπόλεως που θα συνδεθεί με τη γέφυρα αυτή και γιατί αυτό είναι σημαντικό για υποστρατιωτικούς όρους, μα γιατί θα δώσει επιμελητιακή υποστήριξη για τη μετακίνηση, λέω, στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτός ο σταθμός παραγωγής ενέργειας ε, είναι στην Σεβαστούπολη και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν ε, υπήρξε αποκοπή της ενέργειας ε, για την, της Ουκρανίας στην Κρυμαία κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις αντιμετώπισαν πρόβλημα διότι οι στερεωτικές ε, εγκαταστάσεις χρειάζονται διαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως για την Σεβαστούπολη αυτή, αυτή η έλλειψη ας πούμε ήταν πολύ σημαντική. Βεβαίως δεν θα δημιουργηθεί αυτό το, αυτό το κέντρο ε, για να καλύψει τις ανάγκες του αστικού πληθυσμού. Ε, αντιθέτως θα καλύψει τις στρατιωτικές ανάγκες. Ε, φαίνεται να είναι μη αμυντικό, μη στρατιωτικό έργο αλλά στην ουσία είναι στρατιωτικό. Ε, όσον αφορά τη θάλασσα του Αζόφ, σας τα είπα προηγουμένως. Αυτά είναι ουκρανικά πλοία τα οποία θέλουν ε, να, ε, που ανήκουν στον στόλο της Ουκρανίας και θέλουν να ενισχύσουν το στόλο αυτό οι Ουκρανοί. και οπωσδήποτε ξέρουμε ότι η στάση της ε, Ρωσίας δεν θα είναι καθόλου φιλική, αντιθέτως θα είναι επιθετική και πολεμοχαρής. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω εντάχει είναι το εξής. Τον Ιούλιο του 2017 η Ρωσία ε, εισήγαγε ε, κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά και δόγματα όσον αφορά ε, το ναυτικό της πρόγραμμα ε, και την ε, Κρυμαία και την Μαύρη Θάλασσα. Γνωρίζουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη της στρατηγικής η Ρωσία και το ξέρουμε αυτό γιατί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν δύσκολο να κατανοήσει κανείς να προβλέψει την σκέψη της Ρωσίας. Τώρα, δύο ναύαρχοι η Κάσατοφ και Βίτκο και μάλιστα ο ένας από τους δύο ε, ήταν, ε, ε, ο ένας ήταν ο παλαιός αρχηγός των δυνάμεων της Μαύρης Θάλασσας και ο άλλος είναι ο Νίν, επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων, άρα ξέρουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Τον Ιούλιο λέω λοιπόν αυτοί οι δύο ε, ε, ναύαρχοι ε, μίλησαν για την κατάσταση και μάλιστα έδωσαν μία έποψη η οποία κατά πολύ ξεπερνάει την υφιστάμενη κατάσταση. Είπαν λοιπόν ότι η Μαύρη Θάλασσα δεν σταματάει στα γεωγραφικά της ας πούμε περιθώρια αλλά προχωράει στην ουσία, έχει επιπτώσεις πέρα των γεωγραφικών συνόνων της, δίνει δυνατότητα στην ε, για περαιτέρω πρόσβαση προς τα Βαλκάνια αλλά και προς τον Νότο. Εδώ θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. One, next, next, next. Oh, so it's very interesting. I, I did this by myself, but uh, uh, Αυτό το έγραψα μόνος μου ε, αλλά υπάρχει και στην επίσημη ιστοσελίδα ε, της ε, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. σε σχέση με τα περάσματα από τα στενά των Δανελίων. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ η δραστηριότητα είναι η μεγαλύτερη ε, ε, βέβαια η πιο μεγάλη δραστηριότητα ήταν το 73-74 ε, στη διάρκεια εν πάση του Ισραηλο-Αιγυπτιακού της Πριν από πολλά χρόνια είχαμε 94 περάσματα μονάχα το χρόνο αλλά το Νοέμβριο του 2015 βλέπουμε ότι ο αριθμός των περασμάτων έχει ξεπεράσει τα 200 ε, και ε, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να δει κανεί το στοιχείο αυτό για να κατανοήσει την σημασία που αποδίδει στην περιοχή αυτή η Ρωσία. Ταυτόχρονα ε, Βεβαίω είναι σημαντικό, το, τα δαρδανέλια είναι σημαντικό και η δυνατότητα να, περάσματος των δαρδανελίων είναι πολύ σημαντική για την ε, Ρωσία, αλλά και η στάση σε σχέση με την Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν δολοφονήθηκε, όταν ε, σκοτώθηκε ο Ρώσος πρέσβης, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ πολύ κακές σχέσεις με μια πολύ σημαντική χώρα όπως είναι η Τουρκία. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο Ναύαρχος Καστοτόνοφ. Βλέπετε λοιπόν τους γεωπολιτικούς στόχους της Ρωσίας. Τους ανέφερε. Κινείται πέρα από τη σύγχρονη ναυτική ε, στατηγική της ε, Ρωσίας. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να κρατήσουν αντιπαλότητα εκτός της Κρυμαίας και εκτός της βόρειας ακτής του Ευξήνου Πόντου. Διότι αισθάνονται ευάλωτοι, κατανοούν την αδυναμία τους. Ο στόλος τους δεν είναι τόσο σύγχρονος. καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Διαβάζοντας το έγγραφό τους, είναι αρκετά ρεαλιστές. Βλέπουν ωφέλη και μειονεκτήματα της ρωσικής παρουσίας στον Εύξηνο Πόντο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να ανησυχεί κανείς όταν γίνεται ρεαλιστής ο εχθρός του, ο εχθρός και γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Αυτές οι δύο προσωπικότητες ο Ναύαρχος Βίρκο και ο Ναύαρχος Καστοτούανοφ καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω χρόνο. Ναι, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Θα συζητήσουμε μετά, λέει ο Πρόεδρος. Πώς, ποιο είναι το συμπέρασμα. Στο Ατλαντικό Συμβούλιο πρόσφατα αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να πάνε, είπα, να έχουν παρουσία στην Αζωφική θάλασσα. Και ότι εκεί θα συγκεντρώσει τις προκλήσεις της η Ρωσία. Η Ρωσία θεωρεί την περιοχή δική της. Την Αζωφική θάλασσα και τις βόρειες ακτές του Ευξήνου Πόντου. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντισταθμίσει τη ρωσική παρουσία στην Αζωφική θάλασσα και να ασχοληθούμε και με, την, ε, με τον Ουκρανικό στόλο. Τι παρουσιάζει στα προβλήματα που σα ανέφερε, Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Α ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος ε, Πάσκου έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. στρεφόμενος προς το παρελθόν 2014-2015 που ετοιμάζαμε την έκθεση. Προβλέπαμε τότε τις εξελίξεις, τη στατικοποίηση την επόμενη του ευξήνου πόντου. Είχαμε έκρηξη στον Εύξηνο Πόντο μετά τον ψυχρό πόλεμο ήταν χώρος διέλευσης της ενέργειας από κεντρική Ασία προς τους καταναλωτές της Δύσεως. Και λόγω και των δικών του αποθεμάτων, του ευξήνου πόντου. Τώρα ο οικονομικός παράγων επηρεάζεται από τη σατικοποίηση. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς διατηρούμε τα ωφέλη της εκμεταλλεύσεως, της ενεργειακής και της διέλευσης από την περιοχή χωρίς να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την στατικοποίηση. Το παιχνίδι θα κρατήσει πολύ. Υπάρχει ένα στοιχείο όμως για το οποίο θα ήθελα να ξέρω ποια είναι άποψη του πάνελ. Τώρα που οι Ρώσοι έχουν την Κρυμαία, γιατί άραγε αποφάσισαν να κρατήσουν τη Σεβαστούπολη και την υπόλοιπη Κρυμαία ξεχωριστά ε, δικαστικός, νομικός. Ε, έχουμε ομοσπονδία μεταξύ Σεβαστοπόλεως και της υπολείπου Κρυμαίας. Αυτό απαρτίζει την Κρυμαία. Γιατί όσον αφορά την ναυτική παρουσία στον Εύξηνο Πόντο. Εξαρτάται το Μοντρέ και αυτή η κυκλική αναλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η Τουρκία δεν θέλει καν να ακούσει την ιδέα αλλαγής του καθεστώτος αυτού. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμως. Είναι θέμα αρχής. Οι Ρώσοι δεν συμμορφώνονται με τίποτα, με καμία συμφωνία στον αφορά τον έξινο πόντο, Ελσίνκη κλπ. Δεν σεβάστηκαν τίποτα. Όμως σεβόμαστε ακόμα την κυκλική αναλλαγή των δυνάμεων στην περιοχή εμείς. Και σκεφτόμαστε ότι ο τρόπος είναι πραγματικότητα το Μόντρε, άρα δεν το θέτω για τις ναυτικές δυνάμεις. Αναφέρομαι σε άλλα θέματα. Εσείς, κυριέ μου, Αναφερθήκατε στις, στις, στην αεροπορία και κάποιες χερσαίες δυνάμεις. Εντάξει, καλό να κρατήσουμε ανοιχτέ τις γραμμές επικοινωνίας με τη Ρωσία και ένας τρόπος να κρατήσουμε τις γραμμές ανοιχτέ, ένας τρόπος είναι ε, η κυκλική εναλλαγή των δυνάμεων. Ο εκπεριτροπής πλούς. Άρα πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί όσον αφορά την προσέγγιση αυτή και θέλω την άποψή σας. Η Ρωσία και οι Τούρκοι παραδοσιακά είναι αντίπαλοι. Ιστορικός πώς υπήρξαν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι. Αν υπάρχει τώρα μια προσέγγιση, εγώ θα έλεγα ότι οφείλεται αποκλειστικά στην άριστη χημεία μεταξύ των δύο ηγετών της Ρωσίας και της Τουρκίας. Προσωπική χημεία. Αυτό είναι. δεν έχουν σταματήσει να είναι ανταγωνιστέ στην περιοχή. Τώρα αν αυτό αληθεύει ή όχι, βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στετίνα, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη να φορέσετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ που υπήρξατε σαφέστατοι όσον αφορά τη στατιωτική παρουσία στην, στον εύξηνο πόντο. Μέχρι τώρα ακούγαμε κυρίως ποια είναι η ισχύ της Ρωσίας στην περιοχή του Ευξήνου. Μετά Στην Κρυμαία και στη Σεβαστούπολη έχουν μείνει υπολείμματα του στόλου της Ουκρανίας. Ο κ. Στακώστα αναφέρθηκε στην Αζωφική θάλασσα. Η Μαριούπολη είναι ένα πολύ στατικικό σημείο πρόσβασης για πρόσβαση από τον Βορρά προς την Κρυμαία. Έχει απομείνει στόλος εκεί, στον Εύξηνο Πόντο και στην Αζωφική θάλασσα. Υπάρχουν ουκρανικά σκάφη, έχουν απομείνει. Ευχαριστώ κύριε Μπουστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας είμαι ευγνώμων. Άκρους εμπλουτιστικές και ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας. Στην επόμενη σύνοδο κορυφής που επίκειται και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συζητήσεις περί ασφαλείας και αμήνης η νεογέννητη ευρωπαϊκή άμυνα τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να καλύψει όλες τις ανάγκες ασφαλείας της περιοχής. Ξεκινώ από δήλωση που έκανε συναδελφός μου. Αμέσως μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Είπε ή συνάδελφος κάπου Κανείς δεν νοιάζεται για την κατάκτηση της Κρυμαίας. Κανείς δεν θα πεθάνει την Κρυμαία, είπε εκτός από αυτούς που ζουν στην περιοχή, όπως εγώ στη Ρουμανία. διότι πάντα ήταν ιδιαίτερο μέρος ε, για τον επεκτατισμό της Ρωσίας η Κρυμαία. Ιστορικά, μετά τον πόλεμο της Σεβαστουπόλεως, από τα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν ένα ιδιαίτερο σημείο γεωγραφικό για τη Ρωσία. Ερώτηση λοιπόν. Μπορείτε μήπως να μου εξηγήσετε πώς βλέπετε τις σχέσεις μεταξύ της ρωσικής εμπλοκής στη Συρία με το ενδιαφέρον, το συμφέρον που έχουν να ελέγξουν τα στενά. Να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την Ανατολική Μεσόγειο στον Εύξηνο Πόντο. Έχει νόημα είναι μια ε, ε, στρατηγική σφαιρική που ακολουθούν. Μετά, αναφερθήκατε στο ρόλο των ε, στενών, των Δαρδανελίων και τις σχέσεις μελλοντικέ με την Τουρκία. Κάποιοι εδώ στο Κοινοβούλιο λένε ότι πρέπει να αποκόψουμε, να διακόψουμε τελείως σχέσεις με την Τουρκία. Το κατανοώ συναισθηματικός, αλλά στρατηγικός θα είναι καταστροφή διότι θα αφήσουμε τα κλειδιά των Δαρδανελίων εις τα σχήρας του κυρίου Ερδογάν και γιατί όχι του κυρίου Πούτιν. Δεν αναφέρομαι στη μελλοντική πιθανότητα η Ρωσία, η Τουρκία και η Ιράν να απαγορεύσουν πλήρως την πρόσβαση της Ευρώπης προς την Κεντρική Ασία. Αναφέρομαι στην κατάσταση, στο υπαρξιακό πρόβλημα που υφίσταται. Αναφερθήκατε σε προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία της ε, Ρωσίας στον Εύξηνο Πόντο. Τεράστια ρωσική παρουσία. Καλό εσάς, τους επαΐοντες και τους πολιτικούς, να ρίξετε μια ματιά στην πολιτική διαμαρτυρία του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 στο Βουκουρέστι. Εντάξει, διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες κατά κάποιον, ε, κάποιες πολιτικής λογικής. Θα ανακαλύψετε όμως πίσω από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια, τμήματα ευρυδικού πολέμου. Και όταν βλέπετε τα στοιχεία του ευρυδικού πολέμου, επιδάφους ΝΑΤΟ, ίσως εύκολα μαντεύετε ποιοι το διέπραξαν αυτό. Ποιε είναι οι δυνάμεις που αναμειγνύονται και σε σχετισμό μεταξύ Ρωσίας και άλλων εταίρων από την άλλη πλευρά της Ρουμανίας. Γι' αυτό η Ρωσία είναι σημαντική όχι μόνο για τη γειτονική περιοχή, είναι άμεση απειλή, αλλά αντιπροσωπεύει και πρόκληση και πρόβλημα για την ασφάλεια της Ευρώπης εν γέννη. Ή δυνατόν μπορείτε να δώσετε κάποιες λεπτομέρειες Δηλαδή να δούμε γενικά τον εύξηνο πόντο, όπου εκεί, όχι εκεί που οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Ουκρανοί έχουν προβλήματα, όχι συγκεκριμένα σημεία μόνο. Σχολιά σε σχέσεις μεταξύ ευξήνου ε, πόντου και βαλτικής. Διότι τα προβλήματα ασφαλείας είναι αλληλένδετα. Συσχετίζονται. Με τα χαράς λέω σε όλους σας μια και αναφερθήκατε στην ε, πολυεθνική μονάδα στην Κραϊόβα. Υπάρχουν ρουμανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην πολυεθνική μονάδα στην Πολωνία και υπάρχουν Πολωνοί, πολωνικά στατεύματα που ενεργά συμμετέχουν στην ε, μονάδα στη Ρουμανική στην Κραϊόβα. Εδώ βλέπουμε ότι δίδεται μια ευρωπαϊκή απάντηση πρόκληση κατά της ευρωπαϊκής ασφαλείας και εδώ πιθανότατα θα πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Έχω και πολλά άλλα θέματα που θέλω να θέσω, αλλά αληθεύει. Η απάντηση είναι μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ή μέσω των δυνα... δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ που έχει μεγάλη ισχύ και θα αναπτυχθούν συν εξυγχρονισμός των στρατευμάτων των μελών του ΝΑΤΟ, κάτι που κάνουν η Ρουμανία και η Πολωνία αποτελεσματικό τρόπο. Όπως και με αγορά μυντικών συστημάτων από διάφορους προμηθευτές, αλλά δεν μπορούμε να αντιταχθούμε με Κοράνι και βίβλο στην ε, ρωσική ε, επιθετικότητα. Αν το κάνουμε ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο κύριε Μπουστινάρο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στότελμπεργκ, έκανε την επίσκεψη με τους πρεσβευτές ε, και επισκέφθη τα στρατεύματα στην Κραϊόβα το περασμένο Σαββατό και το πέραστο. Ο κύριος Κέλαμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τον κύριο Μποστινάρου και εγώ έχω σχετικά ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική των Ρώσων που έχουν σαν στόχο τη Μέση Ανατολή. Συμφωνούμε, πιστεύω, ότι η κυριαρχία του ευξήνου πόντου δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, στον εύξηνο πόντο αυτό καθεαυτόν, αλλά έχει σκοπό να επεκταθεί στη Μεσόγειο Ρωσία μέσω αυτής προσεγγίσεως. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στατιστικά στοιχεία των ρωσικών πολεμικών πλοίων που διέρχονται τα στενά των δαδανελίων, επίσης και τα στοιχεία για τον εξοπλισμό τους, δυνατότητα εκτοξεύσεως πυράβλων από υποβρύχια κλπ. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και όπως είπε και ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ, ο διάλογος πιστεύω ότι πρέπει να δράζεται επί θέσεως ισχύω και ενότητος. Διότι η Ρωσία είναι εξίσου επικίνδυνη όσο είναι διχασμένη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ε, και διστάζουν να κινηθούν. Αν η σύγκρουση αυτή η διαμάχη μεταξύ βραχυπρόθεσμης ρεαλιστικής πολιτικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, αυτός ο διχασμός να συνεχιστεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Χρειάζεται σφαιρική θεώρηση. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προδιετία για τον εύξηνο πόντο ε, ήταν πολύ επίκαιρο. Και χάρη στον συνάδελφο Πάσκου ε, ισχύει και σήμερα, είναι επίκαιρο. Διότι καταλήγει με μία έκκληση το ψήφισμα. Λέει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κυριαρχήσει, να επικρατήσει επί των ναυτικών και εναερίων δυνάμεων στον εύξηνο πόντο. Αυτό θα ήταν προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ε, ασφαλείας μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από μερικά χρόνια ένας Αμερικανός ερευνητής που εργαζόταν για πολιτική ομάδα προβληματισμού χρησιμοποίησε μια έκφραση που χρησιμοποίησε και πρώην πρόεδρος της Ρουμανίας ο εύξηνος πόντος θα γίνει τελικά ρωσική λίμνη, είπε. Μετά είχαμε την Ουκρανία, ξέρουμε ότι έχουν το στόλο στη Σεβαστούπολη, ε, υπάρχει κίνδυνος η Ουκρανία να αντιμετωπίσει κάποια νέα εισβολή για, για να ισχυροποιηθεί η επικράτηση των Ρώσων στον εύξηνο πόντο. Η γραμματεία δεν βλέπει να ζητά άλλο το λόγο. Θα προσπαθήσω και εγώ να θέσω το δικό μου ερώτημα στα μέλη του πάνελ. Λοιπόν, επί μακρόν προσπαθούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και από πλευράς προκατόχων στην Επιτροπή μας, στην Υποπιτροπή μας προσπαθήσαμε να το θέσουμε το θέμα να συζητηθεί να εξετάσουμε απειλέ εκ νότου και εξ ανατολών και να έχουν προτεραιότητα για τις συζητήσεις μας αυτές οι απειλέ. Βλέποντας τι γίνεται ανατολικά και βόρεια σε αυτή την περιοχή της γειτονιάς μας, φτάνοντας μέχρι την Αρκτική, τι γίνεται στην Βαλτική θάλασσα με στέρηση πρόσβασης στο Καλίνιγκραντ, κάτι που δημιούργησε η Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας και εξοπλισμός, αύξηση του εξοπλισμού, μεταφορά εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας εκεί και επίσης ε, μέσα στατιωτικά για τον έλεγχο της περιοχής και αποκλεισμό της περιοχής για άλλες δυνάμεις και τι γίνεται και στα νότια, στη νότια γειτονιά και τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Ρωσίας, δηλαδή να έχει μία πραγματική παρουσία στη Μεσόγειο προς Νότον. Στα παιδικά μου χρόνια, όταν ήμουν μικρή, είχαμε ένα, παίζαμε ένα παιχνίδι Κάναμε τετραγωνάκια και είχαμε άδεια τετραγωνάκια και προσπαθούσαμε να τα γεμίσουμε. Έτσι ήταν κάπω το παιχνίδι. Να πα από το γεμάτο στάδιο τετράγωνο και το γεμίσει. Να καλύψει το κενό. Η Ρωσία δεν έχει αρκετή οικονομική ισχύ να γεμίσει όλα τα τετραγωνάκια. Δηλαδή να πραγματοποιήσει τα σχέδιά τη. Τι παιχνίδι παίζει. Θέλει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε επιδηματάκια να παίξουμε το παιχνίδι της. Σε κάποια έγγραφα μας λέμε ότι η Βαλτική είναι η πιο ευάλωτη, σε άλλα έγγραφα λέμε ότι ο εύξηνος πόντος είναι ο πιο ευάλωτο. Σίγουρα και τα δύο σημεία είναι ευάλωτα και κυρίως εύξηνος πόντος. Όλος ιδιαιτέρως μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Πάρα πολύ ευάλωτος είναι εύξηνος πόντος. Μακρά ιστορία, ενδεχομένως πάρα πολύ επικίνδυνη. Πώς τα αξιολογείτε αυτό. Σε ποιο βαθμό αυτές οι εξελίξεις είναι πώς να το πω, πώς να το πω, ε, αλλαγές ή πώς πλέκονται, διαπλέκονται όλες οι αλλαγές στην Αρκτική, σε άλλες περιοχές που αναφέραμε. Ε, υπάρχει διασύνδεση Είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι μπλόφα, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν. Στην Ανατολική Ουκρανία βέβαια δεν μπλοφάρουν, ούτε μπλοφάρισαν με την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Αυτά είναι γεγονότα. Όμως δημιουργούν αυτό το κλίμα, αυτή την εικόνα, αυτή την απειλή να επικρέμεται. Ίσως να αποτελεί ένα κομμάτι, πώς να το πω, παραπληροφόρησης. Προσπάθεια παραπληροφόρησης. Βέβαια, είναι γνωστά τα πραγματικά στοιχεία και τα γεγονότα. Θα ήθελα όμως να ξέρω ποια είναι η γενική εικόνα. Όταν μιλάμε για οικονομικές δυνατότητες, αναφερθήκατε στις κυρία για τη στατικοποίηση της οικονομίας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πρέπει να έχουμε επίγνωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται έναντι της δικής μας αφελούς ε, επιχειρηματικότητας της ελεύθερης αγοράς που χρησιμοποιούμε εδώ. Θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Τι σχήματα ακολουθούνται από την άλλη πλευρά. Τι μοντέλα. Όμως, παρόλα αυτά, έχουμε και την ιστορική μας εμπειρία. Βέβαια, είχαμε στατικοποίηση Τη οικονομία κάποιε περιόδους της Σοβιετικής Ενώσεως και δεν λειτουργήσε αυτή η προσέγγιση. Ποτέ δεν δουλεύει αυτό. Μπορεί να το κάνεις αυτό για μια μικρή χρονική περίοδο. Ίσως για να στηρίξεις κάποια δράση. Δεν μπορείς όμως να βασίσεις την οικονομία σου σε τέτοιου μέτρα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας επ' αυτόν κύριοι. Με την ίδια σειρά παρακαλώ. Παρακαλώ αν έχει την καλοσύνη να αναφέρετε την απάντησή σας, να αναφέρεστε στην απάντησή σας στην ερώτηση του Ευρωβουλευτού. Σε ποιον απευθύναστε. Ε, έχουμε περίπου ένα μισάωρο στη διάθεσή μας, 20 λεπτά και κάτι. Παρακαλώ, διαιρέστε το χρόνο ισότιμα. Thank you for some... Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα ερωτήματα και τις σκέψεις σας. Ε, δεν θα μπορούσα μέσα 5 λεπτά να τα απαντήσω όλα όμως παρόλα αυτά. Θα το προσπαθήσω τώρα όσον αφορά τη Ρωσία και την Τουρκία. Ναι, αν υπάρχει κάποια χημεία εκεί μέσα ή όχι. Πιστεύω πως ε, ναι υπάρχει ε, χημεία και ο ε, Πούτιν εκτιμά ηγέτες οι οποίοι μένουν στην εξουσία περισσότερο ε, από ό,τι γίνεται στις παραδοσιακές δημοκρατίες. Γι' αυτό το λόγο εκτιμά τον Ερντογάν για το ότι κατόρθωσε να μείνει τόσο στην εξουσία. Δεύτερον, υπήρξε μια καλή συνεργασία κατά την έναρξη των δύο προεδριών, Πούτιν και Ερντογάν, σε ε, σε αντίθεση με το Κουρδιστάν ας πούμε. Ε, η Ρωσία λοιπόν είχε ε, την διάθεση να εκμεταλλευτεί την, το Κουρδιστάν, από την άλλη οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν την τσετσενία αυτή. Η ανταλλαγή λοιπόν κάπως βελτίωσε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ηγετών, όμως κατά την τελευταία δεκαετία η οικονομία πραγματικά αποτέλεσε την κόλλα, το συνδετικό κρίκο στη σχέση τους. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες Ρώσους στην Τουρκία, οι οποίοι φέρνουν τα χρήματά τους. Υπάρχει εμπορική σχέση με το αέριο, πάρα πολλές ε, ε, εταιρείε κατασκευών της Τουρκίας έχουν επωφεληθεί ε, κατασκευάζοντας στάδια για το επερχόμενο Μουντιάλ. Επίσης ε, υπάρχουν ε, κοινότητες οι οποίες ε, συνεργάζονται για να ενισχύσουν τις σχέσεις. Επίσης μετά το περιστατικό κατάρρευσης του ρωσικού αεροπλάνου έγιναν προσπάθειες επιχειρηματίες, Τούρκοι επιχειρηματίες χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιώσουν τις σχέσεις. Οπότε υπάρχουν ανεπίσημοι δεσμοί οι οποίοι κάνουν τη σχέση αυτή ακόμα πιο ισχυρή. Επίσης, ε, από την άλλη, οι Τούρκοι ε, προσπάθησαν να ε, παίξουν το χαρτί της εξωτερικής πολιτικής. Όταν λοιπόν η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει καλά, τότε η Ρωσία είναι ένας καλός σύμμαχος. Επίσης, η Σύρια ανάγκασε την Τουρκία να στραφεί προς την Ρωσία. Είναι ε, πολύ σημαντικό για αυτούς λοιπόν, ε, λόγω του ότι συνορεύουν ε, με την Σύρια, να συνεργαστούν με την Ρωσία. Δεν χαιρόμαστε για αυτό, δεν χαίρονται για αυτή τη σχέση, αλλά πρέπει να συνεργαστούν. Τώρα όσον αφορά τη Συρία. Αρχικά η Ρωσία προσπάθησε να λύσει στον Κάφκασο τα προβλήματά της με αποτέλεσμα να ανοίξει τις πόρτες για να πούν όλοι οι μαχητές ε, στη Συρία. Αν δούμε τις στατιστικές λοιπόν και τις απώλειες ε, στον Κάφκασο, οι απώλειες έχουν μειωθεί τόσο μεταξύ των αστυνομικών όσο και των απλών πολιτών. και έχουμε ε, το ακόλουθο ε, πρόβλημα. Ε, έχουμε το ISIS και πολλοί θα θελήσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όμως καλό είναι να μείνουν κλειστές οι πόρτες και να μην μπορούν να μπουν στη χώρα. Επίσης υπάρχει η σχέση με τις ΙΠΑ και έχουμε και αυτό το κόμπλεξ της Σοβιετικής Ένωσης τα συναισθήματα υπάρχουν ακόμα εκεί και άμα εξετάσουμε το πώς είναι η ρωσική ηγεσία ε, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι, ε, το τι συμβαίνει. Επίσης ε, είναι και λειτουργικό το σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία. Το θέμα δεν είναι μονάχα ε, το να υπάρχουν ε, βάσεις για επισκευή των πλοίων αλλά και για την κατασκευή ε, πλοίων. Η κατάσταση λοιπόν θα συνεχιστεί και υπήρξε μια ανταλλαγή προσπάθησαν να ενισχύσουν, να προκαλέσουν αυτή την κρίση για να κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο χαλαρή όσον αφορά την Ουκρανία. Προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, όμως αυτή η λογική επικρατούσε. αν κρίνω ε, από τα κριτήρια κυρώσεις υπάρχουν ακόμα, η πρόεδρος παρακαλώ ε, μην ξεκινάτε διάλογο μεταξύ σας, ε, να δοθεί χρόνο σε όλους. Και με ρωτήσατε για τη στρατηγικοποίηση της ρωσικής οικονομίας υπάρχει η πεποίθηση ότι ο στρατικός τομέας της Ρωσίας μπορεί να, είναι, να βοηθήσει την, τον οικονομικό εξυγχρονισμό της Ρωσίας. Υπόθηκε δημοσίως αυτό, όμως ε, δεν ε, μπορούν να γίνουν κάποιες ε, διακηρύσεις, μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες διακηρύσεις για να δούμε το πώς κατανέμονται τα ποσά και αυτό γίνεται βέβαια εις βάρος των κοινωνικών υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της υγείας και άλλων κρατικών δαπανών. Βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα ε, του εξυγχρονισμού μετά από ε, τον πόλεμο με τη Γεωργία, όμως ταυτόχρονα έχουμε ακόμα πιο πολλούς φτωχούς ε, οι οποίοι ζουν, το πώς ζουν με τρία χρόνια μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Για την κυβέρνηση της Ρωσίας όμως είναι σημαντικό να συνεχίσει να επενδύει χρήματα σε αυτό το τομέα διότι πάνω από το 60% των ε, βιομηχανικών παραγωγών στη Ρωσία παράγονται από το στρατικό τομέα και επίσης είναι σημαντικός τομέας και όσον αφορά την απασχόληση. Πρέπει να έχεις να κρατήσεις πιστούς τους πολίτες και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να υπάρχουν συμβόλαια και παραγωγή και ταυτόχρονα χρησιμοποιείται ε, και ως ένα μπραντ ε, καθότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγιάς παγκοσμίω ε, στρατιωτικού εξοπλισμού και με αυτό το λόγο διασφαλίζει την πίστη των πολιτών της Ρωσίας. Δείτε εδώ μπορούμε, παράγουμε, εξάγουμε Ε, ενισχύει την περηφάνεια του λαού καθότι συνεχίζουν να διατηρούν αυτή την παράδοση παραγωγής όπλων. Τώρα όσον αφορά την Ουκρανία δεν έχει ε, μεγάλο ναυτικό ε, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας αλλά και πριν από αυτό δεν ήταν τόσο λειτουργικό το ναυτικό της. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ουκρανία θα πρέπει δυστυχώς να ξεκινήσει σχεδόν από το μηδέν. Ο κίνδυνος είναι ότι ε, καθότι δεν έχει ε, πρόσβαση στη θάλασσα του Αζόφ και εφόσον η Μαριούπολη ε, είναι τόσο ευάλωτη και αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία και έχουμε και την Οδέσα που είναι η τελευταία γραμμή Οδυσσό και εκεί θα πρέπει να ενισχυθεί η στρατιωτική ε, παρουσία, όμως ε, και όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της ε, περιοχής, αλλά και ε, την ε, παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων που θα μπορούν να αποτρέψουν οποιαδήποτε ρωσική ε, επίθεση που δεν βλέπω να γίνει αυτή τη στιγμή καθώς ο στρατός της Ρωσίας δεν είναι ολοκληρωμένος ακόμα. Έχουν λειτουργικές μονάδες και έτοιμες να επιθούν άμεσα όμως δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να διατηρήσουν μεγάλες επιθέσεις. Τώρα όσον αφορά τη Συρία, το, να ανοίξει καινούριο μέτωπο η ε, Ρωσία θα ήταν κάτι τραβηγμένο για τη χώρα. Ο ε, κύριος Χόρελ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ξεκινήσω με ε, μία από τις τελικές ερωτήσεις που μου ετέθησαν. Όσον αφορά τη θάλασσα του Αζόφ, εκεί μπορούμε να, θα μπορούμε να τονίσουμε ότι την στρατιωτική σημασία της Μαριούπολης ως λιμάνι όσον αφορά το ναυτικό ε, της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλισσα, Ε, η Ναυαρχίδα βρισκόταν εκτός ε, του λιμανιού και ήταν το μόνο πλοίο λοιπόν το οποίο δεν ε, κατασχέθηκε ε, μαζί με τους καπετάνιους και το πλήρωμα. Έτσι λοιπόν έχει μονάχα αυτήν την φρεγάτα. Τώρα όσον αφορά τα λοιπά ερωτήματα σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας ε, θέλω να πω ότι είμαι της ε, σχολής ε, ότι υπάρχει μια στρατηγική από την πλευρά του Πούτιν μπορεί να μην είναι καλά οργανωμένο ακόμα στιγμής και όποτε παρουσιάζονται ευκαιρίες της Αδράτη είναι ε, γρήγοροι, ε, δεν ε, αφιερώνουν πολύ χρόνο όπως τη Δύση για να λάβουν μία απόφαση και δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα υβριδικά μέσα τα οποία έχουν και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να είναι αποτελεσματικοί για τους, με τους στόχους τους. Τώρα όσον αφορά την διατήρηση της, του στάτους της μεγάλης δύναμης, αυτό απαιτεί πρώτον να κάνει τις άλλες μεγάλες δυνάμεις ε, να υπαναχωρήσουν, να υποχωρήσει δηλαδή το ΝΑΤΟ, η ΕΠΑ, ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την επιρροή που, ε, δείχνουν, ε, να εκμεταλλευτεί, να δυσχεραίνει μάλλον την συνεργασία που υπάρχει στην Δύση και το βλέπουμε αυτό με τις κυβερνοπληροφορίες που δίνονται Έχουμε επίσης την αντιπαραγωγικότητα ενός ε, ε, βαλτικού μετόπου ε, όπου λέγεται ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τη Ρωσία. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην επιτρέψουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα να προσφέρουν την ευκαιρία την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί η Ρωσία. Ε, σε οποιαδήποτε υβριδικά, περιστατικά δεν θα αποτελούσε έκπληξη για μένα αν ε, βρίσκαμε τη Ρωσία από πίσω. Είχαμε την επιρροή ε, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις δυτικές εκλογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πούτιν προσπαθεί να διασπάσει την δυτική ενότητα και εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα να αποδυναμώσει οποιαδήποτε δυτική χώρα. Επίσης οι σφαίρες επιρροής είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει λοιπόν η Μολδαβία, η Γεωργία και η Ουκρανία να αποτραπεί από το να ε, πάνε πιο ε, δυτικά θέλει να έχει μια γεωπολιτική επιρροή και ε, βλέπουμε να ε, γίνεται όλο αυτό στη Συρία. Δείχνει δηλαδή ότι ε, μπορεί να τα καταφέρει και δείχνει την υποστήριξη στον Ασάντ ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι η Δύση είναι αναποτελεσματική σε μια τέτοια κρίση. Αυτό λοιπόν αποτελεί κέρδος για τον Πούτιν. Τώρα όσον αφορά σε μία από τις ε, διαφάνειες ε, αναφέρθηκε ο ρόλος της ε, Μαύρης Θάλασσας και αυτό θα ήθελα να το τονίσω αποτελεί μία πύλη προς άλλες περιοχές όπου υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι του Πούτιν και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ασκήσει το, τη γεωπολιτική του επιρροή σε αυτό το υπερεθνικό πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε και την Τουρκία που είναι σημαντική για τη Δύση ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ αλλά όχι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι αυτά τα ε, θέματα τα οποία μπορούν, ε, που μπορεί να εκμεταλλευτεί ιδιαιτέρως λόγω της σχέσης που έχουν οι δύο ηγείτες τώρα όσον αφορά το Μοντρό το οποίο το θέμα αυτό αφορά το σεβασμό ε, προς την ε, Τουρκία και αποτελεί λοιπόν μια πρόκληση όλο αυτό ότι ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αυξήσει ακόμα την παρουσία εκεί πέρα, ότι, οπότε για ποιο λόγο αποτελεί εμπόδιο. Εκτός μικροφώνου ο μιλτής. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη Μαύρη Θάλασσα, δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μονάχα ε, σε ε, ναυτικές παρουσίες, ε, θα πρέπει να υπάρχει και παρουσία, κυκλική παρουσία εδάφους και αέρος. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Κουτέλια. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότερες ερωτήσεις απαντήθηκαν. Εγώ όμως θα ξεκινήσω με το τελευταίο σχόλιο, παύρα ερώτηση. Ποιο είναι το παιχνίδι της Ρωσίας ε, και ποια μπορεί να είναι η στρατηγική. Ε, η Ρωσία ε, είναι ε, είναι δύναμη η οποία βασίζεται στο διέρη και βασίλευε ε, και επομένως θεωρούν επίσης ότι οποιαδήποτε δημοκρατική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και προσπαθούν να διαρρήξουν την ε, συνέχειά της και την ενότητά της δεν θα πρέπει να τους ε, επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ε, και ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όπλο μέσω του οποίου κατέρευσε και η, Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, και η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Έχουμε το δόγμα Γερασίμοφ, άλλωστε, το οποίο αναφέρει ότι μπορεί ο έλεγχος ε, να γίνει σε σχέση με την ανάκλαση που μπορεί να έχει ο κίνδυνος ε, ε, σχετικά με, το, με την ομάδα στόχου. Μέσω αυτού προσπαθούμε να επιτύχουμε το βέλτιστο πολιτικό αποτέλεσμα για μας. Αυτό κάνει η Ρωσία χρησιμοποιώντας δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει και η οικονομική οικονομική δυνατότητα, τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Μια άλλη παρατήρηση που μπορώ να κάνω είναι η εξής. Έχω αναλύσει ε, τα έγγραφα της Ρωσίας ε, και βλέπει κανείς και διαπιστώνει ότι το 2020 είναι μια σημαντική ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία ανανέωσης του στόχου, είναι η ημερομηνία αλλαγής διάθρωσης ε, της στρατιωτικής οργάνωσης. Αποτελεί πραγματικά ένα ε, πολύ σημαντικό ε, ε, χρονικό στόχο. Επομένως, για να μπορέσουμε να προβλέψουμε υπάρχουν και να μην τρέχουμε πίσω από εκ των υστέρων, ε, μπορούν να μελετηθούν οι καταστάσεις ε, και βλέποντας ιστορικά την κατάσταση ε, υπάρχει μια εμπειρία σε ένα πολύ ωραίο έγγραφο το NSDP 17 77 μάλλον, του Προέδρου Ρίγκαν. Εδώ, σε αυτό το έγγραφο, αναλύεται η στρατηγική ε, και μπορεί τότε να μιλούσαμε για Σοβιετική Ένωση, αλλά αν διαγράψουμε το Σοβιετική Ένωση και βάλουμε το Ρωσία, μια χαρά ισχύει η στρατηγική αυτή ε, και υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ε, είναι σημαντικά. Είναι αυτή η ηγετική δύναμη και η στρατηγική ηγεσία και στρατηγική λοιπόν ηγεσία η οποία ε, έδωσε την ε, δυνατότητα στην Ρωσία να απλώνεται ε, για να καλύψει τα κενά. Το έκανε και στην Συρία. Τώρα φαντάζομαι ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι πολύ σημαντική. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, την γενικότερη εικόνα. βεβαίω η Μαύρη Θάλασσα σε σχέση με τη Μεσόγειο είναι απαραίτητη στη Ρωσία έτσι ώστε να απλώσει τη δύναμή της μέχρι την ε, Μεσόγειο. Ε, μετά από την προσάρτηση της Κρυμαίας προσπαθεί να δει ε, σε ποια σημεία ε, θα διαραγεί η ενότητα και το μέτωπο ε, έτσι ώστε να μπορέσει να εξαπλώσει ακόμα περισσότερο την δύναμη της Δημιουργεί λοιπόν ε, νέες προκλήσεις μέσω της ε, ε, Μεσανατολής λόγω των τρομοκρατικών απειλών, λόγω των μεταναστευτικών προσφυγικών μάλλον ροών, έτσι ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στη δημοκρατική κοινότητα. Γι' αυτό η Σύνοδος Κορυφής της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των απειλών. Μένει ακόμα δρόμος βέβαια μέχρι την εφαρμογή στρατηγικών που προενεργητικά ε, θα μπορέσουν να ε, ε, αποτελέσουν την απάντηση και στα ευρυδικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει η Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουρκώστα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έγινε μια ερώτηση για το διαχωρισμό κρυμαια Σεβαστοπόλεως. Εγώ μεγάλωσα στην Σεβαστούπολη και ε, όταν ε, ζήσει κανείς, περάσει κάποιο διάστημα χρονικό σε αυτή την πόλη, γίνεται ένθερμος οπαδός της. Και οι κάτοικοι είναι τόσο ε, περήφανοι που είναι μια ειδική περίπτωση Ίσως είναι ε, τόσο περήφανοι και για την πολύ παλιά τους ιστορία. Είναι μακραία η ιστορία της χώρας. Οικοδομήθηκε από τους Έλληνες ε, πριν από πολλούς αιώνες. Και επομένως ακόμα και οι ίδιοι οι Σεβαστοπολίτες δεν θέλουν ε, να θεωρηθούν Κρυμαίοι. Δεν θέλουν να μπουν στο ίδιο καλάθι με τους κατοίκους της Κρυμαίας. και από την πλευρά του Κρεμλίνου το ζήτημα που θέλει να προωθήσει ε, και το Κρεμλίνο είναι ότι η Σεβαστούπολη είναι μια ηρωική πόλη. Τώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς όποιο όρο και όποια ορολογία θέλει μπορεί να, πει, να χρησιμοποιήσει την έκφραση ραπροσμό. Εν πάση περιπτώσει αυτή η προσέγγιση της ε, ε, Τουρκίας και της Ρωσίας μπορεί να αναχθεί στους Ναπολεόντιους πολέμους. Επίσης, ε, Η Τουρκία υπέστη σοβαρά πλήγματα από την πολιτική των πασάδων της ε, Αιγύπτου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρ' όλα αυτά πάντως η Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, επιβίωσε ε, και ο Ατατούρ και ο Λένιν είχαν καλές, ε, καλές σχέσεις. Ε, πριν από αυτό πάντως είχαμε και τη συνθήκη της Λοζάνης ε, που δημιούργησε κάποια ζητήματα. Η Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση προώθησαν κοινές θέσεις σε πολλές περιστάσεις Πάντω, στην παρούσα κατάσταση, η παρούσα κατάσταση μάλλον είναι προ το συμφέρον της Τουρκία να έχει καλε σχέσει ε, με την Ρωσία. Αρχικά, ε, η συνδίκη της ε, Λοζάνη δεν έβρισκε σύμφωνη την Τουρκία, η οποία θεωρούσε τα ύδατα περιών ο λόγο διεθνή. Μετά, από το 1963 πάντως, 1963, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα με την Κύπρο, και επί ψυχρού πολέμου η Ρωσία χρησιμοποίησε κάλλιστα τις αντιδυτικές, ε, το αντιδυτικό αίσθημα της ε, ε, Τουρκίας και μάλιστα είχαμε και στρατηγούς της Ρωσίας που έφτασαν που πήγαν στην Σμύρνη για να συζητήσουν ε, για στρατιωτικά προγράμματα και πρόσφατα μάλιστα είχαμε και μια τέτοια μετακίνηση υψηλόβαθμων ε, στρατιωτικών. Εγώ σας, μιλάω για το 87. Ε, αλλά όλα αυτά σταμάτησαν με την εισβολή στο Αφγανιστάν και η Τουρκία κατάλαβε ότι το συμφέρον της ήταν στο ΝΑΤΟ λόγω της ε, ε, επεκτατικής προς τα νότια πολιτικής της Ρωσίας. Τώρα πάντως οι Τούρκοι δεν αισθάνονται να απειλούνται από την Ρωσία. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Δέστε λίγο τι γίνεται τα τελευταία δέκα χρόνια ε, μεταξύ της Τουρκίας και της Δύσης ας πούμε. Διαρκώς ε, παραπονιέται η Τουρκία ε, γιατί δεν λύνονται, δεν λύνονται προβλήματα ενώ η Ρωσία δίνει βήμα στην Τουρκία μέσω της πλατφόρμας της Αστάνα ας πούμε. That's a main, main aspect, I think. Νομίζω ότι Έκανα το γύρο του προβλήματος και νομίζω ότι δεν έχουμε και χρόνο, πρέπει να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι με αυτές τις τελικές παρατηρήσεις μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ε, ακρόαση η οποία διήρκεσε δύο ολόκληρες ώρες αλλά ήταν τόσο ενδιαφέρουσα όμως. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό να ευχαριστήσω τους ε, τέσσερις έγκριτους ε, ομιλητές μας, ε, καθώς επίσης και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι προφανές ότι θα παραμείνει στο θεματολόγιό μας. Δεν είναι φυσικά η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε για την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τους καλεσμένους μας ομιλητές.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 πρέπει να ακολουθήσουμε την, ε, τη συνήθεια διαδικασία μας και να έχουμε μια ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της ΣΕΝΤΕ uh, ε, στην ε, Trident και στην Νότια και στη Ρώμη και στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ Πρόκειται για δυνάμεις οι οποίες ε, προστατεύουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλαμε να δούμε με ποιο τρόπο το κάνουν, ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έτσι ώστε να μειωθεί η απειλή των ανθρώπων, η απειλή ε, μάλλον να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο, η πληγή των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους ε, στη θάλασσα. Είχαμε λοιπόν ε, μία μικρή αποστολή ΣΕΝΤΕ υπό την δική μου ε, προεδρία. Είχαμε και εκπροσώπους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ο κύριος Εβεμπελέτ. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΛΥΜΠΕ, λοιπόν. Είχαμε επίσης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος ε, Σουλίκα μέλος ε, και της ε, ΣΕΝΤΕ, ε, Λορέντζο Κέζα. Είχαμε εκπρόσωπο της Σικελίας που ήρθε όμως μονάχα στο Σικελικό τμήμα της αποστολής. Αναφέρομαι στον κύριο Σαλβατόρε Ντομένικο Πουλιέζε. Τρεις ήταν οι μέρες της αποστολής, εντός των οποίων καλύψαμε ευρύ φάσμα θεμάτων και πλήθος επιπέδων επαφών με την Ιταλική κυβέρνηση, με διεθνή κέντρα κλπ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μία ενημέρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ιταλίας. Είχαμε λοιπόν μία πάρα πολύ καλή ενημέρωση στο Υπουργείο Άμυνας όπου μας μίλησε ο αναπληκτής υπουργό Άμυνας ε, και είχαμε μαζί του μια ευρεία συζήτηση. Επισκεφθήκαμε επίσης ε, το, στην πράτη Μάρε το αρχηγείο της ακτοφυλακής. Είναι ένα μέρος κοντά στη Ρώμη. και εκεί είχαμε την δυνατότητα να δούμε τις δραστηριότητες του αρχηγείου και να δούμε και τις αποστολές ε, άλλων ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλουν στην ε, προσπάθεια αυτή στα πλαίσια της αποστολής Τρίενα. Επισκεφθήκαμε επίσης και την ε, Ιταλική Βουλή. Το Κοινοβούλιο λοιπόν της Ιταλίας όπου είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων και προσωπικά από τον ίδιο τον Πρόεδρο αλλά και άλλα μέλη πολύ σημαντικά, Πάολα Άλλη πρόεδρο, τον πρόεδρο της ε, ε, Ατλαντικής ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης κλπ. Στη Σικελία τώρα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία επίσκεψη επιτόπου. Ακούσαμε ενημερώσεις από πολλούς ανθρώπους που άμεσα εμπλέκονται με την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Συζητήσαμε με Ιταλούς βέβαια, αλλά και άλλων ε, εκπροσώπους άλλων χωρών, εκπροσώπους της αστυνομίας ε, άλλων κρατών μελών, που βοηθούν την Ιταλική ακτοφυλακή και την ακτοφυλακή γενικότερα. Ενημερωθήκαμε για την αλλαγή των διαδρόμων, την αλλαγή των τρόπων δράσης των διακινητών, γιατί είναι σαφές ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα ε, οι διαδρομές που ακολουθούν οι διακινητές. Πολλά πράγματα μάθαμε. Ε, από την προηγούμενη επίσκεψή μας στην ε, Σοφία, είχαμε, στα, στο αρχηγείο της Σοφίας είχαμε ε, πολλές αλλαγές. Διαπιστώσαμε ότι πολλά έχουν αλλάξει. Ε, και έχουν προκύψει και πολλές αλλαγές ε, μετά από την συμφωνία με την Τουρκία για τον περιορισμό της ροής των μεταναστών στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα σενάρια λοιπόν των διακινητών έχουν αλλάξει και τώρα έχουν εμπλεκεί και Ρώσοι και Ουκρανοί που και αυτοί έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα έχοντας τη βάση τους ε, στο, σε τουρκικό έδαφος. Το θέμα της Λιβύης βέβαια μας απασχόλησε περισσότερο κεντρικό ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις μας. και στην επαφή που είχαμε με το αρχηγείο της ακτοφυλακής στην Βράτικα Μάρε, αλλά και στην επαφή που είχαμε στην ε, Ρώμη με το Κοινοβούλιο, ε, ακριβώς συζητήσαμε το θέμα αυτό και το ίδιο και στην Νάπολη όπου επισκεφθήκαμε το κέντρο ε, κοινών ε, αποστολών ε, στην, του ΝΑΤΟ, κοινών δυνάμεων. Και εκεί το συζητήσαμε, το θέμα αυτό. Και βέβαια είχαμε και μέλη της ε, ε, μέλη της Γραμματείας και είχαμε και μαζί μας και τους ε, συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση αυτή. που είχαμε κυρίως από τον Ναύαρχο Χόλμερ και στο Joint Force Command κάναμε και συζητήσεις για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ the, solving of, of, uh, όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων στη Μεσόγειο όσον αφορά την ε, διάσωση στη θάλασσα σύμφωνα με την ε, Συμφωνία Σάλλας, Σύμβαση Σάλλας. Αλλά συζητήσαμε επίσης και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε ε, να περιοριστεί η ροή, η μεταναστευτική και να μειωθεί λοιπόν το μεταναστευτικό κύμα κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα της Βόρειας Αφρικής και της υποσαχάριας περιφέρειας ε, της ε, Αφρικής, ε, όπου δηλαδή πρέπει εκεί να αντιμετωπίσουμε τα, τις γενεσουεργές αιτίες της μετανάστευσης. Επίσης, συζητήσαμε το θέμα των hot spots Ε, είχαμε την ευκαιρία και να επισκεφθούμε ε, τα κύρια σκάφη της Γιουνάρ Σοφία, αυτά τα οποία συμμετέχουν στις ε, παρούσες επιχειρήσεις. Και εκεί, στο λιμάνι της Μεσίνης, είδαμε και σκάφη τα οποία παρέχονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις για σκοπούς ε, διάσωσης μεταναστών. Μετανάστες οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους ε, λόγω των διακινητών. Βέβαια σε πολλά από αυτά που ακούσαμε, σε πολλές περιπτώσεις και στη Σικελία και στη Ρώμη, ακούσαμε και διαπιστώσαμε ότι οι Ιταλοί ενοχλούνται ε, από αυτό γιατί μπορεί να έχουν όλη την καλή θέληση του κόσμου ε, να ε, συντονίσουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά παρόλα αυτά εδώ μιλάμε για σκάφη τα οποία προχωράνε πάρα πολύ μακριά, φτάνουν σχεδόν στην ακτογραμμή της Λιβύης και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολος ο συντονισμός των σκαφών αυτών και αυτό ενοχλεί τους Ιταλούς. Ήταν πολύ σύντομη ε, η ε, επίσκεψη. Τρεις μόνο ημέρες. Τρεις μέρες όμως κατά τη διάρκεια των οποίων επισκεφτήκαμε τρία πάρα πολύ σημαντικά ε, μέρη. Είχαμε επαφές και συναντήσεις από το χάραμα μέχρι τη νύχτα. Όλα αυτά βέβαια ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Κρίμα που οι, επισκέψεις που μπορούμε να κάνουμε ε, και το μέγεθος της αντιπροσωπείας ε, είναι τόσο περιορισμένο. Μακάρι να μπορούσαν περισσότερα μέλη να συμμετέχουν σε τέτοιες ε, δραστηριότητες. Βέβαια θα σας κάνω και μία ενημέρωση και σχετικά και με την αποστολή του Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, την ετήσια σύνοδο δηλαδή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. αλλά τώρα καλύτερα να σταματήσω την αναφορά μου για την Ιταλία. Yeah. I think there are no questions. It is for the second time I, I speak. Εν πάση περιπτώσει, είναι αργά δεν είμαι και στην καλύτερη φόρμα γιατί ξεκίνησα το ταξίδι μου από τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Όχι, οπότε θα κάνω άμεσα την ενημέρωση σχετικά με την ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, του ΝΑΤΟ. Είχαμε την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λήψη παρουσίας των Προέδρων των αντιπροσωπιών ήμουν εγώ επικεφαλής της αποστολής αυτής. Uh, Εκτός της υποφαινομένης παρίστανται δύο Ρουμάνοι ευρωβουλευτές. Ο κ. Φραντσουλίκα και κυρία Νικολάη. Κατέφθασα Σάββατο. Πέρασα δύο μισή μέρες εκεί. Μαζί με τον κύριο Φραντζουλίκα, που είχε φτάσει προηγουμένως και που είχε συμμετάσχει διάφορες συνεδριάσεις, Ήμουν κι εγώ. Είχαμε ε, ημέρες επιτροπής, ημέρες ολομέλειας και τότε ήρθε η κυρία Ραμόνα Μανέσκου. Ευρωβουλευτήνα του ΕΛΚ από τη Ρουμανία που συμμετείχε και αυτή. Και μαζί με την κυρία Νικολάη μπορέσαμε να καλύψουμε διάφορες επιτροπές και μπορέσαμε να συμμετάσχουμε και στην Ολομέλεια προσπαθώντας να ακούσουμε διάφορες παρουσιάσεις ανάλογα με τον τομέα μας, τον τομέα ενδιαφέροντός μας. Προφανώς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε όλες τις εκδηλώσεις που ήταν σημαντικότατες από την έποψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωκοινοβουλίου. Η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ επεξεργάστηκε και υιοθέτησε 17 ψηφίσματα. Βάση προηγουμένων εκθέσεων. Οι καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές συζητούσαν το θέμα και μετά γινόταν η ψηφοφορία για το κείμενο στην Ολομέλεια. Οι εκθέσεις ήταν πολύ σημαντικές. Υιοθετήθηκε και μια έκθεση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ περί ΝΑΤΟ ε, και συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. καλύφθηκε πολύ έδαφος πιστεύω και λεπτομέρειες. Και διερωτώ με, κατά πόσο οι βουλευτές που ασχολούνται με τον ΝΑΤΟ γνωρίζουν τις λεπτομέρειες ε, όσον αφορά το νομικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όπως τα είδα εγώ τα πράγματα, ήταν αρκετά λεπτόμερης οι εκθέσεις και σε αυτόν τον τομέα και στον τομέα τον ευρωπαϊκό και όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το νομικό περιβάλλον, να το προκαλέσω έτσι. παρουσιάστηκε η μελέτη όσον αφορά τη συνεργασία σε αμυντικά θέματα και τον αρμόδιο φορέα. Ακούστηκαν και κάποιες επιφυλάξεις και τομείς προς ε, συμφωνία μέσω σταδιακών εξελίξεων συζητήθηκαν. Υπήρξε πλήρης ε, υποστήριξη για την έγκριση του ΠΕΣΚΟ. Το ψήφισμα βασίστηκε στην έκθεση του κυρίου Ατήλα Μέστερχάζη είναι Ούγγρος σοσιαλιστής και μέλος της αντιπροσωπείας. παρουσίασε τη θέση του μέσω ψηφίσματος. Ε, Ήταν πολύ σημαντικό το κείμενο. Εστιάστηκε επί του επιμερισμού των ευθυνών και ένας, ένα μέλος της συνελεύσεως από την Λετωνία παρουσίασε το κείμενο που ήταν γνώστης του θέματος. Ο κύριος Κάρινς. Η κοινοβουλευτική συνέλευση επανεξέλεξε τον κύριο Παολάλη ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του ΝΑΤΟ και πέντε αντιπροέδρους και άλλους αξιωματούχους της συνελεύσεως. Είχαμε και σύντομη παρουσίαση της πολωνικής αντιπροσωπείας. Αφορούσε σχέδια για την επικείμενη συνεδρίαση, την, κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ που γίνεται ετησίως Δύο το χρόνο έχουμε. Του χρόνου θα γίνει στη Βαρσοβία. Το πρώτο εξάμεινο. Το Μάιο. Και στο Χάλιφαξ του Καναδά. Το δεύτερο εξάμεινο. Η ομάδα μου γνωρίζει ότι επιλέγεται ο τόπο σύμφωνα με τα σχέδια και τις επιθυμίες τους. Η συνεδρίαση στο Βουκουρέστι ήταν αρκετά σημαντική. Καλήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων. Θεμάτων που αφορούν και τις δικές μας εργασίες και τις τωρινές και μελλοντικές μας αποφάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει κανείς τη συζήτηση. Βέβαια δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου. Ο ρόλος μας εκεί είναι διαφορετικός. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να δούμε τις εργασίες και για μένα που σε πρώτερες θέσεις μου όταν ήμουνα μέλος του Πολωνικού Κοινοβουλίου συμμετείχα ενεργά στις εργασίες της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του ΝΑΤΟ και γι' αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνω σύγκριση τώρα. Το Χάλιφαξ είναι ενδιαφέρουσα από όλοι, αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να συνθέσουμε μια μεγαλύτερη αντιπροσωπεία και μεγαλύτερη αντιπροσωπεία για την ε, συνέλευση την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ εκεί. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για την κυρία Νικολάη και για μένα. Να καλύψουμε όλα τα θέματα που μας αφορούσαν. Ευχαριστώ γι' αυτό την γραμματεία που βοήθησε. Ήταν ικανότατη η γραμματεία ο συνήθως. Είμαστε πολύ καλά χέρια με τη βοήθεια της γραμματείας μας και ευχαριστώ εκ νέου τη γραμματεία για τη βοήθειά της. Ενθαρρύνω τα μέλη να συμμετάσχουν στην αποστολή και να επιλέξουν αυτά τα θέματα, αυτούς τους τομείς. Γιατί είναι σημαντικότατο ζήτημα και για τη μελλοντική μας συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και ΝΑΤΟ. Ε, είναι σημαντική συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Και ενθαρρύνω τα μέλη να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίκολα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ παράκολουσα τις εργασίες της συνέλευσης. Ξεκίνησα Σάββατο πρωί ξεκινάνε πουρνό-πουρνό με τις πολιτικές ομάδες. Ήμασταν μόνο δύο, παρακολούθησα μόνο δύο επίτροπες, γιατί η συνέλευση κάλυψε ε, εγώ την πολιτική ε, επιτροπή παρακολούθησα και της ε, άμυνας. Η Ρωσία συζητήθηκε, η Συρία οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ όσον αφορά δυναμικό και το διαδίκτυο. Πολύ ε, ενδιαφέρον θέμα και συστήνω τους ε, συναδέλφους διαβάσουν στην έκθεση ε, εξοπλισμός της πληροφόρησης. Η Τζεν Κόρντιαν, η Καναδή συνάδελφος ετοίμασε αυτή την έκθεση. Άλλη έκθεση αφορούσε την ασφάλεια στον εύξηνο πόντο. Περιλάμβανε πολύ καλές ιδέες η έκθεση. Συστήνω να παρακολουθείτε τις εργασίες της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του ΝΑΤΟ. Ήμουνα κάπως δυσαρεστημένη, διότι μόνο δύο άτομα δεν ήταν αρκετά, ακόμα και σαν παρατηρητέ που είμαστε, δεν είμαστε μέλη. Η συνέλευση μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε κοντά στους βουλευτές που ασχολούνται με θέματα του ΝΑΤΟ, να μοιραστούμε μαζί τους πληροφορίες και να συνεργαστούμε. πρέπει να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και τη δυνατότητα που έχουμε να εξετάζουμε και να συζητούμε τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, για τα σχόλια. Καταρχά να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πρωτίστως για την συνεργασία. Ευχαριστώ τα μέλη που συμμετείχαν και ενθαρρύνω τους συναδέλφους να συμμετάσχουν. Αξίζει τον κόπο και είναι ευκολότερο να ασκήσει τη δραστηριότητά σου εκεί. Μαθαίνουμε πράγματα εκεί, ενώ διαφορετικά πρέπει να διαβάζουμε για αυτά. Να διαβάζουμε πάρα πολύ τεκμηρίωση. Πολύ δύσκολο να παριστάμε σε επιτροπές βεβαίως και κάθε επιτροπή διεξάγει πολύ καλό έργο, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ συνάδελφοι. Α, ωραία. Λοιπόν, λίγα λεπτά για μια αναδιάταξη και μετά θα ξεκινήσουμε το πολύ ενδιαφέρον επόμενο πάνελ. Θέμα το, το οποίο ήδη το έχουμε συζητήσει. για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων και την ανάλογη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίση, επίσης και θα συζητήσουμε θέματα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ε, συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Ε, περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Παρόλα αυτά, ε, το πρόγραμμα θα είναι αρκετά ενδιαφέρον και αύριο μέχρι τις 12.30 αύριο θα έχουμε το δεύτερο μέρος της συνάντησής μας. Θα ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω ένα θέμα το οποίο ήδη έχει συζητηθεί στη ΣΕΝΤΕ αλλά και σε άλλες ε, επιτροπές και θεσμούς και αμέσως μετά θα περάσουμε ε, στο, στη συζήτηση σχετικά με την συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση πυρηνικών όπλων και την γενικότερη ε, κατάσταση σχετικά με την ε, μη πυρηνική διάδοση. Το θέμα λοιπόν είναι αρκετά μεγάλο. Ε, συζητήθηκε πολύ και γι' αυτό το λόγο δικός μου στόχος ήταν και παραμένει να ξεκινήσουμε την παρουσίαση σε επίπεδο ΣΕΝΤΕ με, ε, ε, με έναν πιο ουδέτερο ε, τρόπο και για αυτό το λόγο επέλεξα, επέλεξα να καλέσω τον κύριο Γιάτσεκ Μπιλίτσα ο οποίος είναι ο κύριος σύμβουλος σε αυτό το ε, περιεχόμενο και ε, και επιπλέον είναι ειδικό απεσταλμένος ε, για ζητήματα μη πυρηνικής διάδοσης και αφοπλισμού και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ήταν ανάμεσά μας δύο φορές και τώρα είναι η τρίτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περίοδου. Ο επόμενος ε, καλεσμένος μας ε, είναι ο κύριος Ρορακίν, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του γραφείου του ΟΗΕ για ειρήνη και ασφάλεια στις Βρυξέλλες. Ασχολείται και ο ίδιος με, την, ε, με τον αφοπλισμό, με ζητήματα αφοπλισμού. Ακολούθως ε, είναι ο κύριος ε, Τόμ Πλάντ, ο οποίος είναι επικεφαλής του προγράμματος του του Ινστιτούτου Ρούση, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο και θα παρουσιάσει το ε, paper του πάνω στο θέμα. Και τελευταίος, αλλά όχι έσκατος, ε, είναι ο κύριος Πάτρικ ε, Κλάουσον ο οποίος είναι επικεφαλής στο Ινστιτούτο Washington, το οποίο βρίσκεται στη Washington και διαχειρίζεται τέτοια ζητήματα. Ε, ύστερα από συζήτηση ε, που θα έχουμε θα ε, ήθελα να δώσω το λόγο αρχικά στον κύριο Γιάτσεκ Πιλίτσα. Παρακαλώ. Uh, members αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτήν ε, τη συνάντηση που αφορά τη νέα ε, συνθήκη του ΟΗΕ αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση σχετικά ε, με την μη πυρηνική διάδοση. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία πάνω σε αυτή τη συνθήκη όπως επίσης και στη συνθήκη απαγόρευσης. Έτσι λοιπόν οτιδήποτε θα πω σήμερα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι δεδομένο. Ε, κάποια στοιχεία σχετικά με τη γενικότερη κατάσταση όσον αφορά την πυρηνική διάδεση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη συνάντηση που, έχει, που είχε στην ε, Γενική Συνάλευση του ΟΗΕ σχετικά ε, με το ζήτημα αυτό. Στην συμφωνία που είχαμε τονίσαμε λοιπόν ότι ο κόσμος ε, πλέον ε, αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση διάζωσης και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η ε, προσοχή μας αλλά και η δράση. Αυτό, σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται δύο ζητήματα. Αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις πυρηνικές δοκιμές και τις δοκιμές πυράβλων από την Βόρεια Κορέα. Οι δράσεις αυτές απειλούν την παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και αποτελούν κατάφορη παραβίαση αποφάσεων ε, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης αποτελούν πρόκληση στο καθεστώς μη πυρηνικής διάδοσης όπως επίσης και τη Συμφωνία Περιμηδιάζωσης ε, για ε, τον ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτή η συνθήκη αποτελεί τη βάση για την μη διάδοση και τη βάση για τον αφοπλισμό. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης αυτής ε, και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ε, εξέλιξη, ανάπτυξη της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη λοιπόν θα προσπαθήσουν τα μάλα για να διασφαλίσουν την επιτυχία αυτή, αυτή της συνθήκης και η πρώτη και δεύτερη ε, Επιτροπή Προετοιμασίας ε, έχουν ως επικεφαλής ε, εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι τελευταίες εξελίξεις στην Κορέα δείχνουν το πόσο σημαντική είναι η συνθήκη περί αποκλεισμού. Αφοπλισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε την υιοθέτηση της απόφασης 2310 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά την κατάσταση στην Κορέα, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν άμεσα κυρώσεις κατά της ε, λαϊκής δημοκρατίας της ε, Κορέας, ε, όπως ορίζεται από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 2375 ε, και επίσης να υπάρξουν και αυτόνομες κυρώσεις ε, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αποπυρηνοποίηση, της, πυρηνικοποίηση της ε, ε, κορεατικής χερσονήσου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη συνεργασία μας με τους εταίρους μας εκεί για την ασφάλειά τους. Ε, ένα άλλο ζήτημα ε, είναι το σχέδιο δράσης το οποίο έχουμε διαπρατευτεί με το Ιράν, το οποίο δείχνει ότι η διπλωματία μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα ακόμα ε, και ε, στις πιο σοβαρές κρίσεις ε, πυρηνικής διάδοσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλες τις πλευρές. Όσον αφορά την προέλευση της νέας συνθήκης, Ε, στην τελευταία συνεδρίαση περιλαμβάνονταν ε, αναφορές στις ανθρωπιστικές συνέπειες οποιασδήποτε, οποιασδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων και παρόλο που το τελευταίο ε, κείμενο δεν ολοκληρώθηκε, τρεις συνελεύσεις διοργανώθηκαν ύστερα από πρωτοβουλία της Νορβηγίας στο Όσλο το Μαρτίο του 2013 Στη συνέχεια με πρωτοβουλία του Μεξικού το Φεβρουάριο του 2014 και από το κράτος μέλος Αυστρίας στη Βιέννη το Δεκέμβριο του 2014 με αυξανόμενη συμμετοχή κρατών αλλά και ΜΚΟ. Η ε, Σύνοδος της Βιέννης είχε ως αποτέλεσμα ε, να υπάρξει ένα ανθρωπιστικό κάλεσμα από την Αυστρία για να συνεργαστεί με, την, με άλλα κράτη-μέλη και την κοινωνία των, ε, των πολιτών για να καλύψει το νομικό κενό και να εξαλείψει τα πυρηνικά όπλα λαμβάνοντας υπόψη τις απαράδεκτες ε, ανθρωπιστικές συνέπειες. Η, ε, γενική, η απόφαση της ε, Γενικής Συνέλευσης που καθιερώθηκε το 2015 ε, προώθησε την, ε, τις διαπραγματεύσεις, τις πολυπερίες διαπραγματεύσεις ε, περί μη διάδοσης και αφοπλισμού. Ενώ το 2016 ακολούθησε ένα συνέδριο το οποίο θα διαπραγματευτεί, θα διαπραγματευόταν ένα εργαλείο δεσμευτικό για την αποτροπή των πυρηνικών όπλων. Μία άλλη απόφαση από την, Ευρωπαϊκή, από την Αυστρία η οποία είχε την υποστήριξη 123 μελών του ΟΗΕ ΕΕ αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 ε, για να γίνει ε, ένα συνέδριο το οποίο ε, θα γινόταν τον Μάρτιο και το Ιούνιο και Ιούλιο φέτος υπό τον πρέσβη Ελέιεν Βέιτ της Κώστα ε, Ρίκα στις 7 Ιουλίου φέτος 122 κράτη υιοθέτησαν ε, με ψήφο που ζητήθηκε από την Ολλανδία το κείμενο μιας ε, συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισαν υπέρ Αυστρία Κύπρος, ε, Μάλτα, Σουηδία και Ιρλανδία. Ένα, ένα το καταψήφισε η Ολλανδία και ενώ τα, η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν συμμετείχαν ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε και στην ψηφοφορία. Η ε, συνθήκη λοιπόν ε, είναι διαθέσιμη προς υπογραφή από την 20 Σεπτεμβρίου του 2017 και μέχρι στιγμής 53 Ίσως οι αριθμοί αυτοί να έχουν αλλάξει όμως μέχρι στιγμής. 53 όμως ε, έχουν υπογράψει μεταξύ αυτών και δύο ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία και η Ιρλανδία. Προσφάτως, στις 6 Οκτωβρίου του 2017, η ε, Επιτροπή ε, Νόμπελ της Νορβηγίας αποφάσισε να απονείμει το βραβείο ειρήνης ε, στην Διεθνή Εκστρατεία Εξάλληψης των Πυρηνικών Όπλων και η δικαιολογία γι' αυτό ήταν ότι η οργανώση αυτή το, παραλαμβάνει το βραβείο αυτό για, την, για το έργο της να αποτρέψει τις καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση πυρηνικών όπλων και για τις προσπάθειές της να επιτύχει μια ε, απαγόρευση με βάση συνθήκη. Θα ήθελα τώρα να σας πω ποιος είναι ο στόχος ε, της ε, συνθήκης. Περιλαμβάνει απαγορεύσεις για την ανάπτυξη δοκιμής παραγωγή ε, αποθήκευση, μεταφορά, χρήση ή απειλή χρήσης ε, πυρηνικών όπλων. Ε, κρατικά μέρη δεν μπορούν να επιτρέψουν αποθήκευση, χρήση πυρηνικών όπλων ή άλλων πυρηνικών εκρηκτικών συσκευών στο έδαφος τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος υπό την δικαιοδοσία τους. Το τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνει μία απαγόρευση για την μεταφορά πυρηνικών πυρηνικών όπλων, όμως κάποια, ε, μέλη ε, θεωρούν ότι με βάση την ερμηνεία του κειμένου το ορίζει κάτι τέτοιο. Ε, κάθε ε, κράτος ε, οφείλει να υποβάλει δήλωση σχετικά αν κατέχει ή ελέγχει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη θα έχουν την υποχρέωση να έχουν δικλείδες ασφαλείες που θα ορίζονται από, την, από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη τα οποία κατέχουν και θα θέλουν να μπουν σε αυτήν την συνθήκη θα πρέπει να εργαστούν για την απόλυτη εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Η ε, συνθήκη επίσης ε, στο άρθρο 6 προβλέπει ε, την ε, βοήθεια των θυμάτων ε, και την προστασία του περιβάλλοντας για άτομα και περιοχές που επηρεάστηκαν από τη δοκιμή των πυρηνικών όπλων. Η βοήθεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το φύλλο και την ηλικία, να παρέχει ιατρική φροντίδα και να βοηθά για την κοινωνική και να είναι κατά του οικονομικού ε, και κοινωνικού αποκλεισμού τους. Ε, ε, θα, οι χώρες αυτές λοιπόν επίσης έχουν υποχρέωση απέναντι σε πολίτες και περιοχές όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτές. Δεν θα πρέπει λοιπόν βάσει του άρθρου 6 να υπάρχουν Διστακμη πάνω σε αυτό. Όσον αφορά ε, σχέση με άλλες συνθήκες, η εφαρμογή αυτή δεν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να, ε, να μην λαμβάνει υπόψη τις άλλες συνθήκες. Ο Γενικός ε, Γραμματέας του ΟΗΕ είναι υπεύθυνο ε, για όλο αυτό. Ε, έχουν εκφραστεί ε, διάφορες απόψεις πάνω σε αυτή ε, την συνθήκη. Από την πλευρά της Αυστρίας, για παράδειγμα, έχει υποθεί ότι το γεγονός ότι τα, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμφωνούν με αυτό δείχνει την διαφωνία που υπάρχει σχετικά με ζητήματα αφοπλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από μέλη μια στρατιωτικής συμμαχίας που προβλέπει έναν ρόλο για τα πυρηνικά όπλα στη στρατηγική της ε, και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τριπλή διαφωνία ε, στην ε, Γενική Συνέλευση σχετικά με τον αφοπλισμό. Ο διαχωρισμός αυτός δεν έχει αλλάξει με τη νέα συνθήκη για την απαγόρευση πυρηνικών όπλων και είναι απίθανο να εξαφανιστεί εκτός και αν υπάρχει μια αλλαγή σχετικά με έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα με έναν αποτελεσματικό και αντικειμενικό στόχο στον οποίο όλα τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν οι διαφορετικές απόψεις αντικατοπτρίζουν λοιπόν την ε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους ε, υποστηρικτές ε, θεωρούν ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα νομικό ε, εργαλείο για την εφαρμογή του άρθρου 6 ε, της συνθήκης. Αυτό απορρίπτεται από ορισμένους και θα ήθελα να ε, σας ε, πω τη δήλωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου ε, την ημέρα που ξεκίνησε, που τέθηκε σε, στη διάθεση προς υπογραφή η συγκεκριμένη συνθήκη. Ε, δεν θα είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο, δεν θα μειώσει τα πυρηνικά οστάσια και ούτε θα ενισχύσει την ασφάλεια καμιάς χώρας, ούτε και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Πράγματι, ε, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε το αντίθετο τη στιγμή ε, που απαιτείται κοινή στάση απέναντι στην διάδοση. Σύμφωνα με τον ΝΑΤΟ, η απαγόρευση έρχεται σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική πολιτική της μη διάδοση και αφοπλισμού ε, θέτει σε κίνδυνο την πρώτη συνθήκη και τις προσπάθειες που γίνονται εδώ και 50 χρόνια για, τον, για τη μη διάδοση και αφοπλισμού. Και επίσης ε, μια νομικ... ένα νομικό σχόλιο από το ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη συνθήκη και γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή από τις χώρες μας όσον αφορά τα ε, πυρηνικά όπλα και γι' αυτό το λόγο δεν θα αποδεχθούμε κανένα επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αντικατοπτρίζει ή συνεισφέρει στην ανάπτυξη ε, εθιμικού διεθνούς δικαίου. Ε, παρόμοιες διακηρύξεις έχουν γίνει από όλα τα ε, κράτη τα οποία έχουν όπλα αλλά και από ε, άλλες χώρες όπως είναι η Ινδία και το Πακιστάν που επίσης διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ε, σύμφωνα με τη Γαλλία τώρα ε, σύμφωνα με μια παρουσίαση που έγινε στις 9 Αυγούστου του 2017 η συγκεκριμένη συνθήκη γύρει τέσσερις κινδύνους ε, που είναι αφενός ε, να, να θέσει σε κίνδυνο τη συνθήκη μη διάδοσης επίσης να θέσει σε κίνδυνο τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας επίσης αποτελεί κίνδυνο για την ευρωατλαντική και διεθνή ασφάλεια Κύρια ε, Πρόεδρε, παρουσίασα λοιπόν τις απόψεις των υποστηρικτών και όσων είναι αντίθετοι ε, σε αυτή τη συνθήκη και τις συνέπειες που έχει. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι δεν υπάρχει μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το ζήτημα και γι' αυτό το λόγο επαφίεται ε, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να αξιολογήσει τις δυνατότητες μιας τέτοιας συνθήκης σε περίπτωση που θα τεθεί σε λειτουργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρεσβευτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόρι Κιν ε, και εκπροσωπεί το Γραφείο Σύνδεσμο των Ηνωμένων Εθνών ε, στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ αξιότιμη Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και τον ειδικό απεσταλμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες του πάνελ. Εκπροσωπώ τη Διεύθυνση Αφοπλισμού του ΟΗΕ παρουσιάζουμε τη συνθήκη για την απαγόρευση ε, των πυρηνικών όπλων. Όπως γνωρίζετε, η συνθήκη εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου Αναστότος έτους. Η σύναψη της συνθήκης είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα. Είναι η πρώτη πολυμερής συνθήκη με συμμετοχή πολλών κρατών που διαπραγματευθήκαμε τα 20 χρόνια. Ξεκίνησε υπογραφές 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τώρα 53 χώρες έχουν υπογράψει. Σωστά είναι τα στοιχεία σας, ειδικέ απεσταλμένα. Και τρεις χώρες έχουν κυρώσει τη συνθήκη η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή που θα έχουν υπογράψει και κυρώσει 50 χώρες. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Βασικές απαγορεύσεις της συνθήκης καλύπτουν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων των πυρηνικών όπλων και συμπληρώνει την αρχιτεκτονική εφοπλισμού και μη διάδοση, κυρίω συνθήκη μη διάδοση και το καθεστώ διαφύλαξη. Αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζεται ότι είναι ακρογωνίω λίθο της γενικής προσέγγισης για μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού τα πυρηνικά όπλα. Η συνθήκη θέτει τα πυρηνικά όπλα στο ίδιο επίπεδο όπως τα χημικά και τα βιολογικά όπλα που το 1925 είχαν θεωρηθεί αυτά σαν ασύμβατα με την αρχή της, ε, του ανθρωπισμού. Η πρόθεση των προδιαγραφών ήταν κάτι πολύ σημαντικό και οδηγούν στην ε, απαγόρευση διάδοση αυτών των όπλων και ίσως και οδηγεί και στην τελική εξάλληψή τους. Η συνθήκη είναι ένα προϊόν της μεγάλης επιθυμίας των περισσότερων χωρών κατών μελών του ΟΗΕ να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον πυρηνικό αφοπλισμό, αντικατοπτρίζει αυξανόμενε ανησυχίε όσον αφορά τον κίνδυνο που δημιουργείται από την συνεχιζόμενη ύπαρξη πυρηνικών όπλων συμπεριλαμβανομένη τη καταστροφική, ανθρωπιστική και περιβαλλοντική συνέπεια που έχει η χρήση του. Επίσης ε, και η απογοήτευση και η πικρία οδήγησε σε αυτό. Οι περισσότερες χώρες είχαν απογοητευτεί για το βαθμό και την κλίμακα του πυρηνικού αφοπλισμού και των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν συμπεριλαμβανών αυτών που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για τη μη διάδοση. Η συνθήκη αντιπροσωπεύει σημαντικό βόμα, βήμα συγγνώμη, και συνεισφορά στην επίτευξη του κοινού στόχου για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα και ελπίζουμε ότι θα αναζωογονήσει, θα δώσει νέα ενέργεια σε προσπάθειες σε παγκόσμια κλίμακα για επίτευξη του σκοπού. Υπάρχουν πολλές δίωδοι για να φτάσουμε σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Όπως ο Γενικός Γραμματέας Γκουτιέρος είπε, η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων θα ενισχύσει προδιαγραφές που είναι κατά των πυρηνικών όπλων Ξεπερνώντα την ανάπτυξη και κατάρτιση αυτών των προδιαγραφών, θέλουμε σφαιρικό διάλογο που συμμετέχουν όλοι ανανεώσιμοι, ανανεωμένη μάλλον διεθνή συνεργασία και πρακτικά μέτρα για μετάκλητη, επαληθεύσιμη και ε, γενικό αφοπλισμό που θα είναι επαληθεύσιμο και σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόρικιν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Διευθυντή ε, του Ινστιτούτου Ρούση, Τόμ Πλάντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα. Ευχαριστώ ε, και τους ε, συναδέλφους εδώ και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών ε, είναι πολύ σημαντικός. Εμείς ε, είμαστε ένα Ινστιτούτο ε, ανεξάρτητο το οποίο αναλαμβάνει στρατηγικές αμυντικές μελέτες και βεβαίως έχει και ένα πρόγραμμα για την διάδοση των πυρηνικών όπλων και την πολιτική σε σχέση με αυτό του οποίου ηγούμε. Οπωσδήποτε δεν εκφράζεται εδώ η θέση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασίλειου. Στο Ινστιτούτο έχουμε πολλά προγράμματα, μεταξύ των οποίων ε, και το θέμα ε, της μη διάδοσης, ε, της απαγόρευσης διάδοσης των πυρηνικών όπλων, της σταθεροποίησης κλπ. Θα ήθελα να αναφερθώ ενδεχομένως λίγο πιο διεξοδικά σε θέματα τα οποία έθιξαν οι προηγούμενοι ομιλητές όσον αφορά την συνθήκη και ίσως να πω και κάποια πρακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει ακολουθήσει ο Γενικός Γραμματέα Γουτιέρες. Επίσης, θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σε δύο περιπτώσεις ε, ε, απαγόρευσης ε, διάδοσης αναφέρθηκε και ο, ο, ο σύμβουλος πρέσβης στο θέμα αυτό ε, σε σχέση με την ε, ε, σε σχετικά με την Κορέα και βεβαίως να συγχαρούμε και την Άικαν για αυτό που έχουν κάνει γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουν κάνει μεγάλη εκστρατεία όσον αφορά το θέμα αυτό όσον αφορά την αξιολόγηση της συνθήκης εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο αντίκτυπος της συνθήκης θα είναι ε, σημαντικός. Ε, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, συν, ε, λένε ότι αυτή η συνθήκη είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, συνθήκες και ότι οπωσδήποτε θα ε, συμβάλλει στην απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Βεβαίως υπάρχει και μία σχετική ασάφεια, το είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένω. αναφέρθηκαν μάλλον στα σημεία στα οποία η αναφορά είναι λεπτομερής. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία όπου οι είναι ασαφής. Πρώτον, ε, σχέση ανάμεσα ε, στη σύμβαση και την απαγόρευση ε, διάδοσης των πυρηνικών Νομίζω ε, ότι είναι πάρα πολύ, είναι πιο εύκολο να δούμε τις πολιτικές ενδεχόμενες επιπτώσεις, αλλά όχι ε, τόσο εύκολο να προγράψουμε τις ε, δικαστικές ενδεχομένως, νομικές μάλλον επιπτώσεις. Εγώ είμαι δικηγόρος, ασχολούμαι με διεθνές δίκαιο, αλλά και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρίς την δημιουργία νομικών υποχρεώσεων για τους προσυπογράφοντες. Αυτή η συνθήκη δηλαδή θα πρέπει ε, να δημιουργεί νομικές ε, υποχρεώσεις. Ε, αυτή η σύμβαση, η συνθήκη, συγγνώμη, NPT, θα πρέπει να λάβει υπόψη την, κυρίως την αδυνατότητα εφαρμογής της, κυρίως από τις χώρες οι οποίες διαθέτουν ήδη πυρηνικό όπλο. Επίσης, η κεντρικότητα και η κεντρική σημασία του NPT ε, θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Παρεμβάσεις ε, ε, πολλών χωρών στις προπαρασκευαστικές εργασίες της συνθήκης για την απαγόρευση πυρηνικών όπλων και την κατάσταση των πυρηνικών όπλων μας έδειξε ήδη τον δρόμο επίσης στη συνθήκη υπάρχουν και κάποιες ε, νομικές αντιφάσεις ε, ωστόσο, δεν πιστεύω ότι οι, εκ, οι απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν στις προπαρασκευές εργασίες αντιπροσωπεύουν όλες τις ε, χώρες. Ε, και αν ήμουν στη θέση σας, εγώ θα παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο θέλω να δούμε από κοντά, είναι το θέμα της της εξακρίβωσης. Ε, εδώ ε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και τις, τα όσα έχουν λάβει χώρα ιστορικά σχετικά με την αξιολόγηση του οπλοστασίου του Σαντάμ Χουσεΐν και του Ιράν και από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα ε, να υπάρξουν επιβεβαιώσεις ε, σωστές και ε, επιβεβαιωμένες. Ε, οι συνολικές συμφωνίες για τα μέτρα, για αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, οι safeguards, ε, μπορεί να διασφαλίσει μονάχα ότι ε, είναι σωστή η συνθήκη, αλλά όχι απαραίτητη και ισχύουσα. Είναι κρίμα που η συνθήκη δεν έχει αδράξει αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε να κάνει το πρωτόκολλο υποχρεωτικό και αναφερόμενος δηλαδή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο ε, σε αυτό το οποίο θέτει το άρθρο 6. Η διαπραγμάτευση ε, ε, του, της συνθήκης στο σύνολό της, αλλά ιδιαίτερος του άρθρου 6, έδειξε ότι υπάρχουν και στην Νότια Αφρική, στο Ιράκ και τη Λιβύη πυρηνικά προγράμματα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα. Η περίπτωση του, της, και της Νότιας Αφρικής έδωσε την, μάλλον κατέστησε επαφή, την ανάγκη να υπάρξει ε, από πιο κοντά ε, ανάλυση των θεμάτων ε, και μελέτη όλων των εγγράφων τα οποία νομίμως ή όχι έφτασαν στα χέρια της υπηρεσίας. Βεβαίως τώρα μέσω των conferences των διαφόρων εμπλεκομένων μελών μπορούν να λυθούν και να προωθηθούν ενημέρων, επιμέρους προβλήματα. Το θέμα είναι οι ελεγχόμενες χώρες θα συμμετέχουν υπάρχουν ε, στις, ε, στην επιβεβαίωση. Αυτό δεν έχει λυθεί. Τρίτον, θέματα ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ε, η συνθήκη έτσι όπως έχει γραφτεί ε, δίνει την ε, δυνατότητα σε ε, όλες τις χώρες να αντιμετωπίσουν το θέμα και να έχουν κυρώσεις. Ειδικά δίνει τη δυνατότητα στις χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά όπλα. Ενδεχομένως όμως κάποιες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ανάλογα με την χώρια στρατηγική τους ίσως και χώρες όπως η Σουηδία που είναι αλλά όχι μέλος του ΝΑΤΟ ε, να τους, ε, να βάλει σε μια θέση η οποία ενδεχομένως δεν θα είναι τόσο ευνοϊκή. Επίσης, ε, όσον αφορά τις καλές πρακτικές, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως ας πούμε η επίπτωση που μπορεί να έχει σε ελεύθερες χώρες οι οποίες έχουν, ελεύθερες δημοκρατικές χώρες οι οποίες κατέχουν το πυρηνικό όπλο. Ε, η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν, η Βόρεια ε, Κορέα αλλά και η Ινδία έκαναν ε, ε, πολλές δραστηριότητες lobbying και άσκησης πίεσης και ενδεχομένως εκεί να μην έχει η κοινωνία των πολιτών και τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θέματα αυτά. Το ζήτημα είναι να δούμε, να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αντιμετωπιστεί το θέμα των πυρηνικών ε, ως γενικότερη απειλή της ε, ε, ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από όλες τα αρνητικά στοιχεία ή τις αμφιβολίες τις οποίες εκφράσασα, ε, οπωσδήποτε η συνθήκη αυτή μπορεί να είναι ικανοποιητική ε, όσον αφορά την απαγόρευση πυρηνικών έπλων και την κατάσταση των πυρηνικών όπλων. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες οι οποίες έχουν τα πυρηνικά όπλα, και ε, ε, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, κυρίως όσον αφορά το σκέλος των απειλών στην ε, ασφάλεια. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου να θυμηθούμε ότι ε, ε, και οι θέσει των δύο πλευρών μπορεί να είναι ε, θεμιτές Γι' αυτό λοιπόν ζητώ, κάνω έκκληση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να βρει τρόπους έτσι ώστε οι δύο πλευρές να μπορέσουν να συζητήσουν και να εκθέσουν τα, τις αρχές τους η καθεμία. Ε, στο προήμιο της ε, συνθήκης ε, αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και οι διαδικασίες επιβεβαίωσης θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες. Για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν πυρηνικά αναγνωρίζονται, αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει τα κύρια σημεία εμπλοκής να αντιμετωπιστούν ένα προς ένα. Ας πούμε στην ε, η κατάσταση στην Ινδία, η Βόρεια Κορέα, ε, η Ρωσία, η Κορέα η οποία είναι εκτός οποιασδήποτε συνθήκης. Μήπως θα μπορούσατε να ε. μιλάτε λίγο πιο αργά γιατί είναι αδύνατο να διερμηνεύσουν οι διερμηνείς. Ναι, με, με ενθουσιάζουν τόσο πολύ αυτά τα θέματα που δεν μπορώ να συγκρατηθώ, λέει ο μιλητής. Θα τα ξαναπώ λοιπόν, θα συνεχίσω ε, πιο αργά. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χώρες οι οποίες δεν κατέχουν τα πυρηνικά όπλα ε, να μπορέσουν να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Η Ινδία, ο το Πακιστάν, η Ρωσία η οποία βασίζεται στις πυρηνικές δάμεις, η Βόρεια Κορέα η οποία βρίσκεται εκτός της αρχιτεκτονικής της μη διάδοσης. Είναι ορισμένες από, από τα, ορισμένα τμήματα της διεθνής ε, κοινότητας που θα πρέπει να ε, ληφθούν ε, υπόψη και που θα πρέπει να που μπορούν να αποτελέσουν και εύκολους στόχους της διαδικασίας lobbying. Αν έχω χρόνο, θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια για το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Πρώτο σημείο. Θα σας πω κάτι παραφρασμένο,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 δεν, ε, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να δούμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση στο Ιράν. Ε, σχεδόν ε, όλες οι περιπτώσεις εμπλουτισμένου ουρανίου, ουρανίου έχουν μελετηθεί για τη χώρα αυτή. 25 χρόνια διαπραγματεύσεων και συγκεκριμένης μελέτης δεν έδωσαν και καλά, τόσο καλά αποτελέσματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς τώρα ελπίζουν όλοι ότι ε, θα μπορέσουν να προωθήσουν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Εγώ το 2011 όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά ήδη μου έλεγαν τα ίδια πράγματα. Όσον αφορά τώρα την συμμόρφωση ε, του ε, ουρανίου και τα συμπεράσματα της, της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες ο Καναδάς για να επιτύχει το πρότυπο της ε, υπηρεσίας ε, χρειάστηκε πέντε χρόνια. Επομένως, οπωσδήποτε ε, και για την περίπτωση του Ιράν θα περιμένουμε τουλάχιστον πέντε χρόνια, όχι περισσότερο. Ε, και όταν ε, ε, λέμε ότι δεσμεύεται το Ιράν, εννοούμε ότι δεσμεύεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες. Όσον αφορά τη λαϊκή δημοκρατία της Βόρειας Κορέας, μπορώ να πω απλά ότι υπάρχουν, υπάρχει κίνδυνος ε, να, η Βόρεια Κορέα να αναπτύξει ε, το, το πυρηνικό της οπλοστάσιο ε, μόνη της από τη στιγμή που λείπει οποιαδήποτε διπλωματική διεργασία. Ε, πιστεύω ότι εδώ υπάρχει ένας ε, συγκεκριμένος κίνδυνος, ότι η Βόρεια Κορέα δηλαδή ε, θα διαφοροποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο μια και δεν θα διαθέτει όλα τα στοιχεία και θα κάνουν ε, λοιπόν ε, τα δικά τους ε, πυρηνικά με τις δικές τους δικλείδες ασφαλείας. Αν ξεκινήσει μια κλιμάκωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθεί. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξει σαφώς στους στους συμμάχους της ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτεί ε, τέτοιες θέσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάτρικ Κλάουσον από το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε να παραστώ. Να τονίσω ότι αυτά που λέω σήμερα είναι προσωπικές απόψεις, δεν εκπροσωπώ κάποιον. Η συνθήκη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων είναι αξιέπαινο στόχο. Στόχο που ετέθη το 1947 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όταν η κυβέρνηση αμερικανική προσεφέρθη να αποσυρθεί από το πυρηνικό τη μονοπόλιο και να παραδώσει τα πυρηνικά όπλα στον ΟΗΕ. Δυστυχώ όμω είχε αντίρρηση έντονη η Σοβιετική Ένωση γιατί ανέπτυσε δικό τη οπλοστάσιο. Ο ίδιο στόχο προευλήθη από τι ΗΠΑ το 1986 όταν ο πρόεδρο Ρόναλντ Ρέγκαν στη Σύνοδο Κορυφή του Ρέκιαβικ ε, πρότεινε στον πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τη Σοβιετική Ενώσεω να παραιτηθούν δύο χώρε στο πυρηνικό πλωστάσιο και δυστυχώ η Σοβιετική Ένωση δεν δέχτηκε αυτή την προσφορά. Όμω σήμερα αυτή η συνθήκη για απαγόρευση νομίζω ότι ε, κάπως είναι παραπλανά από πιο αποτελεσματικού τρόπους να πετύχει στο στόχο και τελικά καθυστερεί από την επίτευξη των στόχων που θέτει. Παραπλανεί εγώ θα έλεγα διότι το σύστημα μη διάδοσης έχει αποτελματωθεί τα τελευταία χρόνια ε, και θα πρέπει να προχωρήσουμε, να βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε. Πρόσφατα είδαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το κοινό σχέδιο δράσεως, JCPOA είναι τα αρχικά του, και αυτή η συμφωνία προσέφερε πολύ σημαντική πρόοδο και μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτή και να προοδεύσει. Και ελπίζω, σαν διεθνής κοινότη, να μπορέσουμε να αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας, ούτω ώστε να σημειωθεί ιδέουσα προόδο με βάση αυτή τη συμφωνία. Και τελικά να καταλήξουμε σε γενική μόνιμη πρόοδο σε όλο τον κόσμο, παρά να μην περιορίσει την περίπτωση του Ιράν και να είναι χρονικά περιορισμένη λύση. Τι έκανε αυτή η συμφωνία που δεν την προσωμιώνουμε με τις συμφωνίες που έχει πετύχει η Διεθνής ε, Οργάνωση Νομικής Ενέργειας, ε, προσφέρει διάφορους τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Να παραθέσω κάποιους τομείς. Πρώτον, οι εγκαταστάσεις πυρηνικές του Ιράν ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο. Στις περισσότερες συμφωνίες οι διεθνείς η υπηρεσία ατομικής ενέργειας εξαρτάται από επιθεωρητές που πάνε κάθε δύο μήνες και συλλέγουν εγγραφές από τις μονάδες που παρακολουθούνται. Υπάρχει μια τεχνολογία της δεκαετίας του 60 όταν διαπραγματευόμασταν τις συνθήκες και είναι ξεπερασμένες τεχνολογίες. Τα πάντα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο σήμερα. Αυτή η διαφορά σημαίνει διαφορά διμήνου όσον αφορά τον εντοπισμό παρεκκλήσεων. Δεύτερον, και τίθενται και όρια όσον αφορά τη χρήση ε, εμπλουτισμένου ουρανίου σε χαμηλό βαθμό εμπλουτισμένο που μπορεί να έχει στα χέρια του το Ιράν. Άρα, έχουμε σοβαρό περιορισμό όσον αφορά την ταχύτητα με τον οποίο το Ιράν μπορεί να παράξει το σχάσιμο υλικό. Άρα, μπορούμε να βασιστούμε υπάρχει αποθήκη στο Καζακστάν με, το προϊόν και να θαρρύνουμε και άλλες χώρες να δεχθούν την αρχή σύμφωνα την οποία περιορίζεται το ποσό του, χαμηλ, του εμπλουτισμένου ουρανίου σε χαμηλό βαθμό εμπλουτισμένου που μπορούν να έχουν στα χέρια τους. Και μετά έχουμε όρια πόσο μπορεί να εμπλουτιστεί το ουράνιο, τίθενται ανώτατα όρια, άρα Μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο μια χώρα προχωρά σε επίπεδα ε, εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι εμπλουτισμένο σε βαθμό που μπορεί να παράξει πυρηνικά όπλα. Επίσης έχουμε και ένα άλλο στοιχείο του πυρηνικού καυσίμου που μένει εκτός ε, που δεν ελεγχόταν από την Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας αποτελείται yellow cake, είναι μια ουσία Επίσης ελέγχουμε και τα ορυχεία και τις μονάδες επεξεργασίας των ορυκτών Αυτά παλιά δεν ελεγχόταν, τώρα ελέγχονται με αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει κάτι άλλο. Και οι μονάδες ε, κεντροφυγικού ή επεξεργασία ε, πρέπει να ελέγχονται επίσης. Αυτό δεν γινόταν στο παρελθόν. Και προβλέπεται και χρονοδιάγραμμα για ε, πρόσβαση σε αδήλωτε τοποθεσίες και εγκαταστάσεις κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται τα συμφωνίες του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας. Αυτά τα στοιχεία της συμφωνίας του Ιράν είναι στοιχεία που σιγά σιγά θα απομακρυνθούν και το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να τηρήσει αυτές τις συνιστώσεις μετά την εκπνοή ε, του χρονικού ορίου που καθορίζει τη συμφωνία. Και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να ενθαρρυνθούν και άλλες χώρες να εθετήσουν πανεφερή μέτρα. Καλύτερο θα ήταν να, να αφοσιώσουμε το χρόνο μας και την προσπάθεια να εφαρμοστούν τα μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα και μόνιμα. Έτσι θα πετύχουμε καλύτερα τους στόχους να μειώσουμε την απειλή του πυρηνικού πολέμου από τη μια συμφωνία αγόρευσης. Όπως σας είπα, ξεγελάει παραπλανά αυτή η συμφωνία απαγόρευσης και είναι και ένα εμπόδιο. Γιατί, πρώτα απ' όλα, μια τέτοια συμφωνία απαγόρευσης μπορεί να είναι επιβλαβή για τη φήμη των συμφωνιών ελέγχου των όπλων. Ο προλαλή σα αναφέρθηκε ε, στο σύμφωνο Κερόκ Πριάντ του 1928 όπου τα συμβαλόμενα μέρη θεωρούν ότι είναι ο πόλεμο σαν ένα μέρο εθνική πολιτική σε σχέσεις με άλλη χώρα και η λύση όλων των διευθετήσεων ποτέ δεν θα πρέπει να επιδιώχεται παρά μόνο με ειρηνικού τρόπου. Αυτό το σύμφωνο του 1928 υπεγράφει από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και άλλε 30 χώρε, πάνω από 30 χώρε. Αυτή η συμφωνία δεν είχε κανένα αντίκτυπο και ξέσπασε ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από κάποια χρόνια και τι έκανε να βλάψει τη συμφωνία συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών για την επόμενη τριακονταετία. Θεωρήθηκε ότι τροφοδοτεί ε, υποκριτές δικτάτος αυτή η συμφωνία ενώ οι πιο τίμοι υποχωρούσαν. Θα ήταν ατυχές αν αυτή η συνθήκη είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τις συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών. Μειώνει την εξοπιστία τους, άρα μειώνεται και η υποστήριξη που τους ε, παρέχεται. Ε, δεύτερον, η συνθήκη δεν καλύπτει τα βασικό πρόβλημα, τα βασικά προβλήματα που εμφανιστήκαν και τονιστήκαν το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν όσον αφορά την εξάλληψη των πυρηνικών όπλων από πλευράς χωρών που δεν έχουν τα όπλα ακόμα. Το Ιράν ήθελε να αναπτύξει δυνατότητα να έχει πυρηνικό όπλο και αυτό είναι διαφορετικό από τα πυρηνικά όπλα. Τι ήθελε το Ιράν, να είναι σε θέση να παράξει πυρηνικά όπλα γρήγορα και δεν μπορούσε να του σταματήσει η φυστάμενη συνθήκη. Λίγα μπορούσε να κάνει για τη μη διάδοση. Τεράστιο κενό δημιουργείται. Α δούμε το πρόγραμμα του Πακιστάν, το πυρηνικό. Το 1984, Ο AQ Khan, σημαντική προσωπικότητα τότε στο πρόγραμμα, έγραψε στον πρόεδρο Ζία Ουλχάκ του Πακιστάν και είπε ότι θα μπορούσε να ε, κατασκευάσει βόμβα αν ήθελε. Δεν ανέπτυξε, δεν κατασκεύασε τη βόμβα λόγω ε, μια νομοθεσία των ΙΠΑ που έλεγε ότι θα σταματήσει η βοήθεια από Αμερική προς το Πακιστάν αν το Πακιστάν κατασκεύασε πυρηνικό όπλο. Τι έκανε το Πακιστάν που έχει γίνει γενικά αποδεκτό. Συναρμολογούσε βόμβες και άφηνε μια βίδα ξεβίδωτη. Έτσι είχαν πει μυστικέ υπηρεσίε των ΗΠΑ για να εξηγήσουν τι κάνει το Πακιστάν. Δηλαδή οι βόμβες αυτές ήταν έτοιμες εκτός από ένα κομματάκι. Έλειπε ένα κομματάκι που πρέπει να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί. Άρα, είχε είναι η δυνατότητα να έχει κανείς ένα όπλο ατομικό σε τέτοια προχωρημένο στάδιο και η σύμβαση δεν το καλύπτει. Αυτή η σύμβαση τα κάλυπτε και τις είπα. Τι θα μπορούσαν να κάνουν είπα. να αποσυναρμογήσουν τα όπλα τους, να αφήσουν τα κομμάτια των όπλων αποθηκευμένα σε ένα μέρος να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι να συναρμολογούν γρήγορα ξανά τα όπλα και μετά αυτή η χώρα θα ήταν σε θέση να ετοιμάσει δεκάδες πυρηνικά όπλα μέσα σε λίγες μέρες και εκατοντάδες πυρηνικά όπλα σε εβδομάδες. Και αν θεωρείτε ότι οι χώρες που δεν έχουν πυρηνικά όπλα θα το κάνουν αυτό, εντυπωσιάζομαι από την αισιοδοξία σας. Δηλαδή αυτή η συνθήκη μας αφήνει σε μια κατάσταση που είναι πολύ κοντά στην κατάσταση τη σημερινή. Κάνει ελάχιστη διαφορά όσον αφορά τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που υπάρχουν στην πράξη στον κόσμο. Μας κάνει αισθανόμαστε όμως ωραία, αλλά στην πράξη δεν έχουμε αποτέλεσμα και θα μπορούσε να θαρρυνθούν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν παρόμοια κατεύθυνση, να κάνουν το κόλπο του Πακιστάν, ανακοινώνοντας ότι συμμορφώνονται ακόμα με την ε, συνθήκη. Λοιπόν, πρέπει να ανησυχούμε και κυρίως για τη Μέση Ανατολή, αυτό που μελετώ, να, να ανησυχούμε για το Ιράν από τη στιγμή που λήξουν οι περιορισμοί προβλέπονται από το κοινό σχέδιο δράσης, όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, τότε το Ιράν σε ένα μήνα θα έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είναι καλή κατάσταση. Καλύτερα προσπαθήσουμε τους περιορισμούς αυτούς να τους κάνουμε μόνιμους και καθολικού περιορισμού αυτούς τη Συμφωνία του Ιράν. Να μην πάμε προς συνθήκη, που η συνθήκη επιτρέπει στα κράτη να είναι μια στροφή της βίδας ε, πέρα, πιο μακριά από το να έχουν στα χέρια τους έτοιμη μια πυρηνική βόμβα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω ε, το ε, λόγο στα μέλη, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική δήλωση ως πρόεδρος. Αρχικά θα ήθελα να επαναλάβω ε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου ε, για τον ΟΙΕ Πήρα το ρίσκο πριν από μερικές εβδομάδες να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση στη ΣΕΝΤΑ γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα που έχει, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις ε, μεταξύ των κρατών μελών και με προσοχή αποφάσισα να παρουσιάσω διαφορετικές απόψεις ε, και απόψεις ειδικών πάνω σε αυτό Ε, φέρνοντας και έναν εκπρόσωπο του ΟΗΕ και τώρα μετά από αυτή την παρουσίαση ευελπιστώ να μπορείτε να δείτε την πολυπλοκότητα αυτού του θέματος ε, και ελπίζω επίσης ε, να καταλαβαίνετε για ποιο λόγο αποφάσισα να μην καλέσω τους νίκητες του Νόμπελ Ειρήνης διότι οι ε, κάμερες ή ε, τα ΜΜΕ ε, και η παρουσία αυτών δεν βοηθά στην αξιολόγηση αυτού του θέματος. Είμαστε νομοθέτες και βέβαια είμαστε πολιτικοί όμως ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά ζητήματα είμαστε ε, η γέφυρα ε, που ενώνει τα κράτη μας ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία εκτιμούμε σαν έναν οργανισμό που συνεισφέρει στην παγκόσμια ειρήνη. Θα πρέπει λοιπόν όμως να είμαστε υπεύθυνοι και γι' αυτό το λόγο έλαβα την απόφαση αυτή. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Στάντζο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω αυτά που μόλις είπατε. Νομίζω ότι για να γίνουν, να διεξαχθούν ειρηνικά ε, οι ε, εργασίες μας έπρεπε να είναι έτσι. Εδώ ακούσαμε ε, πολλά πολλές ακαδημαϊκές τοποθετήσεις για θέματα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά εδώ δεν είμαστε για να δεχτούμε αυτήν την δημοσιότητα όσο και αν είναι σωστό το ε, θέμα και οι προσπάθειες ε, που καταβάλει κάποιος. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ ακούμε πολλά και πολλές απατηλές έτσι, ιδέες, ψευδεστήσεις κατά κάποιο τρόπο. Ε, από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι καθόλου καλό, είναι καταστροφικό και σας, καταστροφικό και σας εξηγώ γιατί το θέμα των πυρηνικών ε, στις διεθνείς σχέσεις ποιο είναι, είναι η διάδοση η οποία ενισχύεται. Και αυτή η ε, συνθήκη δεν θα σταματήσει τη διάδοση των πυρηνικών. Αυτό είναι γεγονός. Ένα δεύτερο ενισχυτικό γεγονός είναι αυτή η αμφισημία η οποία υπάρχει στα πυρηνικά δόγματα πολλών χωρών όσον αφορά τη μείωση του κατοφλίου. Οι Ρώσοι, οι Πακιστανοί, ε, είναι πυρηνικές δυνάμεις οι οποίες αφήνουν μάλλον καθαρά να εννοηθεί ότι ε, η προσφυγή στα ε, πυρηνικά δεν θα αφορούσε μονάχα την παραδοσιακή αποτροπή αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μια κίνηση ε, ε, η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει τη συμβατική παρέμβαση ή τέλος πάντων ένα μείγμα ανάμεσα στη συμβατική και πυρηνική παρέμβαση. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ρεαλιστικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επομένω, οι καλές προθέσεις, τα καλά αισθήματα, η τέλο στόχη συνολικής, ε, συνολικού αφοπλισμού, πολύ καλά είναι και πυρηνικη παρεμβαση αυτα ειναι τα θεματα τα οποια ρεαλιστικα πρεπει να αντιμετωπισουμε επομενω οι καλε προθεσει τα καλα αισθηματα οι υψηλη στόχοι συνολικου αφοπλισμου πολυ καλα ειναι και ομορφα αλλα περνούν ξιστά από το στόχο, δεν βρίσκουν στόχο. Ε, πολύ συνετά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ε, καλεί ε, να ακολουθηθεί μια λογική πρακτική οδός αλλά η πρακτική οδός δεν είναι η ιδεολογική τοποθέτηση που πρέπει να έχει μια συνθήκη όσο και αν έχει γενναιόδορους στόχους. Ε, στην ουσία ο, η πρακτική οδός είναι ε, τα μέτρα εμπιστοσύνης τα οποία δεν αποφασίζονται μέσω διαταγμάτων και συμβάσεων συνθήκων αλλά οικοδομούνται. Επομένως, ε, αυτή η συνθήκη ε, ε, μπορεί να είναι γενναιόδορη, τη χαιρετίζουμε, τη θεωρούμε σωστή, καλή κτλ. Αλλά δεν πιάνει το στόχο της και το θέμα είναι ότι δημιουργούμε ψευδεστήσεις στην κοινή γνώμη των ε, δυτικών κρατών, ε, εκεί που έχουμε ε, ιδιαίτερα στιβαρούς μηχανισμούς, έχουμε κοινή γνώμη η οποία ενδιαφέρεται, ενώ έχουμε χώρες οι οποίες κατέχουν την, την πυρηνική βόμβα και όμως δεν πρόκειται να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες ευαισθητοποίησης της κοινή τους γνώμης. Εδώ δείχνουμε ένα είδος αφέλειας, μία ακόμα φορά δηλαδή, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της ετερογένειας ενδεχομένως της, ε, των θέσεων που έχουν και πραγματικά θεωρώ ότι πολλές είναι οι χώρες οι οποίες με πολύ μεγάλη αφέλεια αντιμετωπίζουν και υποδέχονται αυτήν την συνθήκη ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή δόγματος και τη μείωση του κατοφλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, που ε, μου δώσατε το λόγο ε, και για το γεγονός ότι οργανώνεται αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι λοιπόν λένε και τονίζουν επίσης, γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο θέμα, ε, πόσο ε, μεγάλη απειλή αποτελούν για την ανθρωπότητα τα ε, πυρηνικά όπλα. Επίσης υπόθηκε ότι ότι υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την απαγόρευση, όμως όλο αυτό δεν αποφέρει τίποτα. Όσον αφορά τη λογική αυτή δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω ε, το πώς, ε, για παράδειγμα, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα χωρίς να, επιστρέψουμε, να επιτρέψουμε και το άλλο. Γιατί λοιπόν θα πρέπει αυτή η συνθήκη απαγόρευσης να έρχεται σε αντίθεση με τη συνθήκη NPG ε, έτσι ε, λοιπόν, αν το υπογράψω αυτό σήμερα, τότε πώς θα, υπογράφονται, πώς θα απαγορεύονται άλλες απαγορεύσεις. Ε, με βάση τη λογική το θεωρώ ανόητο λοιπόν. Ε, μπορούμε να κάνουμε το ένα επιτρέποντας και το άλλο. Μπορούμε να ακολουθούμε συγκεκριμένους στόχους και οι στόχοι αυτοί έχουν συγκεκριμένα βήματα. Ακόμα και στο NPT, λοιπόν, ο στόχος ε, ο τελικός στόχος ε, της, ε, του αφοπλισμού δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να, να συμμετάσχουμε σε αυτό. Οι πυρηνικές δυνάμεις και το ΝΑΤΟ με εξαίρεση την Ολλανδία δεν συμμετείχαν καθόλου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσαν να επηρεάσουν ε, το κείμενο, το χρονοδιάγραμμα, να ε, επηρεάσουν ε, ποια σημεία του NPT θα κρατήσουμε, ποιες, ποιοι κανονισμοί μετάβασης θα υπάρχουν, όμως καθόλου δεν συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν καμία διάθεση ποτέ ε, δεν σκοπεύουν ποτέ να γίνουν μέλη αυτής της ε, συνθήκης. Ε, αν αυτό λοιπόν έγινε πριν τις διαπραγματεύσεις, εάν υπόθηκε τόσο ξεκάθαρα, τότε ε, προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω την προσπάθεια για κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα εν τέλει ε, αφορά να μην καταλήψουμε ε, τους στρατηγικούς στόχους των πυρηνικών όπλων δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε την ε, εναλλακτική της πρώτης κίνησης. Ε, είπατε εσείς, Τανζόν, ότι, ε, ότι είναι αφελής όλοι αυτοί, όμως εγώ θεωρώ θεωρώ αυτήν την προσέγγιση πέρα ως πέρα επικίνδυνη. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία δεν αποδέχομαι Έχω επίσης το ερώτημα αυτό το ε, πάντα πώς θα αξιολογηθεί και Ποιος λοιπόν είναι ε, εν τέλει ο αφελής, εμείς που συζητάμε για αυτό. Ε, η Επιτροπή του Νόμπελ είναι αφελής, ο ΙΕ είναι αφελής. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται άλλο πια να συνεννοούμαστε για τέτοια ε, πράγματα, γι' αυτό το λόγο θα σας ε, παρακαλούσω να επικεντρωθούμε στην σημασία της μη διάδοση, ένα ζήτημα το, για το οποίο διαδήλωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ποιο λοιπόν θα είναι το μέλλον για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μποτίλβα λεγό. Θα ήθελα και εγώ να ε, συγχαρώ ε, την ε, ομάδα που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, όμως παρόλα αυτά δεν συμφωνώ με την πρόεδρο για ποιο λόγο δεν μπορούμε να τους έχουμε μαζί μας. Όμως αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, θα ήθελα ε, να απευθυνθώ στον κύριο Μπιλίτσα, ο οποίος λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέση για αυτό. Ίσως η Κομισιόν και το Συμβούλιο όμως εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε υιοθετήσει ε, μία θέση στις 27 Οκτωβρίου του 2016 λάβαμε μία απόφαση σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση όπου χαιρετήσαμε το έργο το οποίο είχε γίνει ως τότε στον ΟΗΕ για να μπορέσει να διαπραγματευτεί ένα δεσμευτικό οργαλείο για την απεργόρευση των πυρηνικών όπλων και έχει στόχο την πλήρη απαγόρευση αυτών. Αυτό είχε γίνει τον Οκτώβριο και επίσης καλέσαμε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό το έργο. Ο τελευταίος ομιλητής λοιπόν είπε ότι ακόμα κι αν, το, ε, ε, εγκρίναμε αυτή τη συνθήκη και την υπογράφαμε δεν θα είχε ε, σημασία, δεν θα σήμαινε κάτι ε, αναρωτιέμαι λοιπόν για ποιο λόγο, εάν η Σουηδία το σκέφτεται αυτό, για ποιο λόγο έχουμε τέτοια πίεση από τη ΣΥΠΑ και από το ΝΑΤΟ να μην υπογράψουμε και αυτό ε, επηρεάζει και αμφισβητεί όλη τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Σουηδίας ε, και των χωρών του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούμε να έχουμε κοινέ στρατιωτικέ ασκήσεις. Αν αυτή η απαγόρευση λοιπόν εν τέλει δεν σημαίνει τίποτα, τότε δεν υπάρχει και λίγο, λόγος ε, ώστε το ΝΑΤΟ και οι ΙΠΑ να προσπαθούν ε, να πιέσουν ε, την ε, σουηδική κυβέρνηση να μην υπογράψει. Και επίσης υπόθηκε ότι είναι θέμα το οποίο συζητάμε. Αν περαστεί από το Σουηδικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε αξιολόγηση αντιτύπου, να εξετάσουμε τι συμβαίνει με αυτό. Ε, γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι περίεργο ε, το γεγονό ότι εφόσον δεν σημαίνει τίποτα, ε, για ποιο λόγο να μην το αφήσουμε. Δεν μπορώ να μείνω και να ακούσω τις απαντήσεις που θα δώσετε ε, διότι έπρεπε ήδη να βρίσκομαι σε μια άλλη συνάντηση. Θα ήθελα όμως να πω ότι εφόσον έχουμε αυτή την συνθήκη σημαίνει ότι το NPT δεν έχει λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά όσο πιστεύαμε και γι' αυτό το λόγο απαιτείται ένα επόμενο βήμα και ε, δεν αισθάνομαι ότι είναι πολύ σύγχρονο. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι από τις υπήρους ε, που ε, δεν θα πρέπει να είναι από τις υπήρους που δεν το παίρνουν σοβαρά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Αυτές οι παρουσιάσεις ήταν άκρως ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την αναλυτική προσέγγιση που ακολουθήσατε για το θέμα. Ανεξάρτητα από τους διάφορους εορτασμούς θα πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα με σοβαρότητα και ξέρουμε ότι στις διεθνείς συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο πάντα ε, καταλήγουμε σε αυτή την κατάσταση. Για κάποιους φορείς του δυτικού κόσμου κάθε διεθνή συμφωνία γίνεται και εσωτερική νομοθεσία της χώρας καμιά φορά ε, εντάσσεται στο συνταγματικό δίκαιο. Η περισχή του απλού δικαίου είναι νομικά δεσμευτικό. Έχουμε πλουραλισμό στην Ευρώπη. Οπότε οι διεθνείς νόμοι ε, αναφέρονται και χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές και εφαρμόζονται πράγματι οι διατάξεις των συνθήκων και των νόμων. Αν έχουμε κάποιες άλλες χώρες τους αντιπάλους μας, αυτοί τι κάνουν. Είναι πολιτικά εργαλεία αυτές οι διατάξεις για τις αρχές. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Χρήσιμο από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται για να εφαρμόζονται κάποιες πολιτικές. Άρα δεν έχουμε συμμετρία, αλλά έχουμε το φαινόμενο του καθρέφτη. Έχουμε λοιπόν αυτές τις συμφωνίες που μας δεσμεύουν εμάς, μας δένουν τα χέρια και έχουμε από τη μία αυτούς και τους άλλους από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιούν αυτά τα έγγραφα, αυτές τις συμφωνίες για να δέσουν τα χέρια μας. Όσον αφορά εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πυρηνικά όπλα είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι μια πρόκληση. Διότι πιστεύω ότι όλοι, όλοι μας, αλλά ιδίως κάποιες συγκεκριμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν κάποιο περιφερειακό γείτονα. Ή όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικές έχουν έναν άμεσο γείτονα, ο οποίος στο δόγμα του περιπολέμου και στις πρακτικές δραστηριότητε του έχει κάνει κάτι το οποίο αποτελούσε πολιτική χρήση των απειλών περί ε, χρήσεως των πυρηνικών όπλων. Υπάρχει μακρά περίοδος κυρώσεως για αυτή τη συνθήκη. Αν τίποτα δεν συμβεί, δεν αλλάξει, εντάξει καλώς, θα αλλάξει η κατάσταση. Στο πολεμικό δόγμα της Ρωσίας διαβάζουμε περί τακτικού πυρηνικού χτυπήματος. και κάποιες φωνές το λένε ξεκάθαρα. Αναφέρονται σε τακτικά πυρηνικά πλήγματα. Ας θυμηθούμε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Είπε ότι σε αντίπεινα οι ΙΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα για να αντισταθούν ή να απαντήσουν σε κάποιο πυρηνικό πλήγμα που δέχτηκαν. Και όσον αφορά τη Ρωσία, σε περίπτωση σύραξης που θεωρεί ότι είναι σύγκρουση ή κάποια ένταση και η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει νικά όπλα. Λοιπόν, η Λιδία Λίθος για αυτό το έγγραφο ποια είναι, να δούμε κατά πόσο αλλάζει την καθεστική ατάξη ή όχι. Δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα αυτή τη χρονική στιγμή. Η Σαμπίνε Λόζιν ανέφερε και αυτή την αφέλεια. Είμαστε αφελείς και δεν θα έπρεπε. Και αυτές οι διεθνείς συμφωνίες δεν θα πρέπει να αφορούν κάποιο όραμα του κόσμου ή να χρησιμοποιούνται για λόγους πολιτικής προπαγάνδας, ακόμα και αν είναι ειρηνική αυτή η προπαγάνδα. Θα πρέπει να είναι η πολιτική μας αυτή, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ειρήνη. Και γι' αυτό όλοι είμαστε διστακτικοί και προβληματισμένοι αυτή η NPT, η συνθήκη μη διάδοση των Πυρηνικών όπλων, δεν λειτουργεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο είναι εικονικό και το οποίο δεν είναι πρακτικό να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για τις απαντήσεις. Παρακαλώ όμως αν έχετε την καλοσύνη, διακεκριμένα μέλη του πάνελ, να είστε σύντομοι, διότι ίσως να έχουμε προβλήματα με τη διερμηνία που πρέπει να τελειώσει την ώρα της. Λοιπόν, με την ίδια σειρά. Ο κύριος Μπελίτσα, πρέσβης. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα θέματα. Θέση ισχύ και κάποιες αποσαφηνήσεις. Θυμάμαι ότι ε, τίθεται σε ισχύ 90 μέρες μετά την πεντηκοστή ε, επικύρωση. Ε, άρα δεν γίνεται αυτόματα. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας κάνει έκκληση για αφοπλισμό. Νομίζω ότι αυτός ο όρος αφοπλισμός, αφοπλισμό που μπορεί να σώσει ζωές, κάτι τέτοιο πρέπει να είπε, πάμε καλά. Και εσείς το ερμηνεύσατε ως ε, ε, ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα και για, πιο μικρά όπλα, ε, για μικρό οπλισμό όπως τα ελαφρά όπλα ας πούμε. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά την ε, αναφορά ότι δεν ε, δουλεύει, δεν λειτουργεί καλά η συνθήκη, η παλιά συνθήκη. Είναι μια συνθήκη όμως η οποία ε, λειτουργήσε μέχρι ένα μεγάλο βαθμό όσον αφορά την μη διάβευση και είναι σαφής η θέση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτή τη νέα συνθήκη, την NPT. Ε, επίσης βεβαίως ξέρουμε τι, το περσινό ψήφισμα ε, γιατί εκεί περιλαμβάνονται και κάποια στοιχεία ε, τα οποία επιπροσθέτως ε, αναφέρονται στην, ε, στον αφοπλισμό και τη μη διάδοση. Ε, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορούμε να μιλήσουμε μονάχα για συμφωνημένη θέση και συμφωνημένη θέση είναι μόνο αυτή ε, η οποία έχει περάσει από την ομόφωνη θέση των χωρών, από τα συμβούλια, διορθώνω από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κτλ. Είμαι αρκετά πεπισμένος ότι δεν αναφέρεται ε, η αναγνώριση των πυρηνικών στην, ε, στην περιγραφή της αποστολής μας. Ο κύριος Ρόρι Κίν, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα σχόλιά τους. Ίσως και εγώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο, είναι επίγον να βρούμε ε, τρόπους ε, για να ε, διαγράψουμε τα πυρηνικά από τον ε, κόσμο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω όλοι και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ξέρουμε ότι επίσης ότι δεν έχουμε ενιαία θέση και η συνθήκη η απαγόρευσης το λέει και το δείχνει από την άλλη πλευρά, όπως είπε και ο βουλευτής, είναι σημαντικό να βρούμε ε, νέους τρόπους ε, διαλόγου, έτσι ώστε με το καινοτόμο τρόπο να προχωρήσουμε, κυρίως με τις χώρες οι οποίες έχουν ε, πυρηνικά. Αυτές έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη να πάρουν ενεργό μέρος στην αναθεώρηση της πτυγιού ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ε, του κόσμου. Το δεύτερο ε, ζήτημα το οποίο ανεφέρθη είναι ποια είναι τα στοιχεία ε, τα οποία διαφοροποιούν την συνθήκη απαγόρευσης από τη συνθήκη για την μη διάδοση. Η συνθήκη για την μη διάδοση υποστηρίζει και για την απαγόρευση υποστηρίζει και ολοκληρώνει κατά κάποιο τρόπο τη συνθήκη για την μη διάδοση και αυτό αναφέρεται και στο προήμιο και σε πολλές διατάξεις. Ε, ε, το αφήγημα ότι δήθεν υπάρχει διάσταση νομίζω ότι μπορεί να δώσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πλάν. Κοιτάξτε, θα ήθελα να μην απαντήσω άμεσα, αλλά να σχολιάσω τα όσα υπόθηκαν. Λοιπόν, κάπου, ε, κύριε Ταμσόν, κάπου, κάπου λησμονήσαμε. Μιλήσατε για αντικείμενες ε, απόψεις. Από την αρχή των συζητήσεων του 2010 παρακολουθώ τις που δεν έχουν μεταβληθεί. Τι επαναλαμβάνω, ότι ο διάλογος κινείται με τρόπους όπου και οι δύο πλευρές και υπάρχουν πλευρές μπορούν να συνεργαστούν επί συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου πυρηνική χρήση, χρήση πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρέ μπορούν να συμφωνήσουν ότι είναι προαπαιτούμενο για να πάμε προ την εξάλληψη των πυρηνικών ε, όπλων. Μερικά πράγματα να πω, δάτω μου ευκαιρία να μιλήσω μετά τον συνάδελφο για να απαντήσω ξανά σε αυτά που μίλησαν για την σύγκριση τη συνθήκη απαγόρευση και τη συμφωνία ε, διάδοση των πυρηνικών όπλων. Σε είναι άποψη των περισσότερων χωρών, όχι μόνο το ΙΕ, όχι όλων. Άρα, όταν θα σε ισχύει η συνθήκη, που θα γίνει γρήγορα, θα ξεκαθαριστούν αφισβητούμενες, ε, τα αφισβητούμενα σημεία. Έτσι θα καθησυχάσουν κάποιες ανησυχίες, αυτές που περιέγραψα κι εγώ και έτσι αντιμετωπιστούν και κάποια τα προβλήματα που ανέφερε η κυρία Λόζινγκ. Αν δικαιολογείται να περιγραφόμεθα ως αφελής, τότε θα λυθεί αυτό το θέμα. Δεύτερο κρίσιμο για τη διάσκεψη. Πού εστιαζόμεθα. Ποιες χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα. Υπόκεινται στην δράση κοινότητας οι φιλελεύθερες χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, εκείνες που μπλοκάρουν ε, τον αφοπλισμό αλλού, ε, Πακιστάν και η διάσκεψη για τον αφοπλισμό κλπ. Είναι ένα συγκεκριμένο πρακτικό βήμα μπορούν να κάνουν οι χώρες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις επικρίσεις που ακούγονται. Ευχαριστώ. Ο κ. Κλάρσον. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα για να λειτουργήσει μια απαγόρευση είναι η εξακρίβωση. Αν δεν λυθεί αυτό, η απαγόρευση δεν θα είναι βιώσιμη. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα εξακρίβωσης Πώ αποφεύγει αυτό το πρόβλημα που είπα, που έχουν αποσυναρμολογήσει τα όπλα του κάποιε χώρε και μπορούν γρήγορα να τα συναρμολογήσουν. Ήμουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμετείχα σε πάρα πολλέ συζητήσει για το πόσο θα χρειαστεί η Ιαπωνία να παράξει ένα μεγάλο πλωστάσιο πυρηνικών όπλων ε, πάνω στου ε, πυράβλου. Και έτσι που έχει προγραμματίσει το πρόγραμμά τη το διαστημικό και του πυρηνικού και πυρηνική ενέργεια η Ιαπωνία ήταν πολύ καλά σχεδιασμένα για να μπορεί να γίνει ο συνδυασμό των δύο γρήγορα. Η απάντηση σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ είναι ότι η Ιαπωνία θα χρειαστεί μήνε και όχι πολλού μήνε για να έχει χιλιάδους, ε, μια χι, ε, περίπου χίλιου διπυρωτικού πυράβλου με πυρηνική κεφαλή. Αυτό δεν είναι καθησυχαστικό, άμα σκέφτεσαι την απαγόρευση. Αν μια χώρα όπω η Ιαπωνία έχει αυτού του είδου τη δυνατότητα. Άρα πρέπει αυτό το πρόβλημα να το καλύψουμε αν θέλουμε να λειτουργήσει η απαγόρευση. Και είναι ένα παράδειγμα των περίπλοκων προβλημάτων που πολλέ ώρε είχα περάσει όταν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, προβληματιζόμενο, επεξεργαζόμενο και δεν τα λύσαμε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι στου βασικού λόγου για του οποίου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο προ το στόχο που έχουμε θέσει από μακρόν επί 70 χρόνια να απαλλαχθούμε από τα πυρηνικά όπλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ εργάζεται άκρο να σταματήσει τη συνθήκη. Δεν γνωρίζω. Διότι νομίζω ότι η συνθήκη κάνει και πολλά. Αλλά νομίζω ότι ανησυχεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, θεωρεί ότι η συνθήκη θα είναι ένα βήμα, πρώτο βήμα σε μια διαδικασία και ανησυχούν για τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ήρθε το τέλος αυτού του σημείου της ημερησίας διατάξεως, αλλά και των σημερινών συζητήσεων. Ολόκληρη ημέρα, εξαντλητική, άκρος ενδιαφέρουσα, Ευχαριστώ το διακεκριμένα μέλη ε, του πάνελ. Παρακαλώ χειροκροτήστε και εσείς μαζί μου. Ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση. Αύριο ξεκινάμε στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.